Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, βουλευτές της Επιτροπής ε, ΑΦΚΟ, τις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω, να καλωσορίσω και τους βουλευτές ε, της Συνδεδεμένης Επιτροπής της Επιτροπής Απασχόλησης και να θυμίσω ότι οι Επιτροπές Ρέτζι, Γιούρι και ΦΑΜ έχουν και εκείνες προσκληθεί σε αυτήν εδώ την ακρόαση. Να καλωσορίσω την Ντομπράφκα Σουίκα, αντιπρόεδρο που ορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Αρμόδια για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία. Να θυμίσω ότι η Ντομπράφκα είναι συνάδελφός μας εδώ και χρόνια και πάντοτε με χαροποιεί όταν ένας υποψήφιος ή μία υποψήφια επίτροπος προέρχεται από τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θεωρώ πως είναι κάτι θετικό, γιατί έτσι ε, θα σημαίνει πως θα έχουμε ακόμα πιο θετικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και την παρακολούθηση των δεσμεύσεων που αναλύθηκαν στη διάρκεια της ακρόασης, να θυμίσω ότι ο ε, σκοπός της ακρόασης είναι να αξιολογήσουμε τις γενικές ικανότητες, την ευρωπαϊκή προσήλωση και την προσωπική ανεξαρτησία της υποψήφιας αντιπροέδρου, καθώς και τις γνώσεις της για το μελλοντικό της χαρτοφυλάκιο, καθώς και τις ικανότητες κοινωνιακές της ικανότητες. Θυμίζω ότι προβλέπεται η μεσιαναμετάδοση των ακροάσεων από το site του Κοινοβουλίου που θα είναι δυνατόν κανείς να προχωρήσει και στην μαγνητοσκόπησή τους. Να σα θυμίσω επίση ότι η Επιτροπή Γιούρη αφού εξέτασε την δήλωση οικονομικών συμφερόντων της, αντιπροε... της αντιπροέδρου δεν διαπίστωσε ε, και δεν ε, έκανε καμία αντίρρηση στην ε, διεξαγωγή αυτής εδώ της ακρόασης. Η υποψήφια αντιπρόεδρος θα κληθεί να κάνει μια προφορική δήλωση εναρκτήρια και στη διάρκεια της ακρόασης θα ε, υποβληθούν 25 ερωτήσεις που θα διαιρούνται σε μπλοκ 25 ε, λεπτών εκάστη. Επερώτηση θα μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά από την απάντηση της Αντιπροέδρου για τη διάρκεια του πενταλέπτου. Θα είναι λοιπόν ένα λεπτό για την υποβολή της ερώτησης από πλευράς του κάθε βουλευτή, δύο λεπτά για την απάντηση της, αντι... της υποψηφίας αντιπρόεδρου με τη δυνατότητα ε, συμπληρωματικής ερώτησης ή επερώτησης από τον ίδιο βουλευτή για όχι πάνω από ένα λεπτό και μια απάντηση ενός λεπτού επίσης για την από πλευράς της υποψήφιας ε, ε, αντιπροέδρου. Στο τέλος η υποψήφια αντιπρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια τελική δήλωση όχι πάνω από 5 λεπτά. Να σας θυμίσω επίσης ότι το βιογραφικό σημείωμα της υποψηφίας Πρόεδρου και οι απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις έχουν διανεμηθεί σε όλους τους βουλευτές και έχουν δημοσιευθεί και στο site του Κοινοβουλίου. Η ακρόαση θα διαρκέσει τρεις ώρες, δηλαδή μέχρι τις 9.30. Ε, θα θυμίζω ότι η υποψήφια την Πρόεδρος έχει υποδείξει ότι θέλει να κάνει συζήτηση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την έννοια, τη δομή, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο της διάσκεψης για το μέλλον της ε, Ευρώπης επί τη βάση του concept paper που θα υποβάλει ως σημείο εκκίνησης αυτής της ίδιας ε, συζήτησης. Εγώ εύχομαι η υποψήφια Πρόεδρο να μπορέσει να μας πει κάποιες από τις σκέψει της για αυτό το θέμα στη διάρκεια αυτής εδώ της ακρόασης. Διότι για την ε, Επιτροπή μας ε, η διάσκεψη, η συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης ε, έχει θεμελιώδη σημασία. Να θυμίσω στην Αντιπρόεδρο πως ήδη έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης από πλευράς της Επιτροπής μας το θέμα αυτό και η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών ε, είπε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπηθεί με κατάλληλο τρόπο να μπορέσει να έχει ενεργό ρόλο και να υποβάλει προτάσεις επί τη βάση των εργασιών που έχουν γίνει ήδη στην προηγούμενη θητεία. Όλοι οι βουλευτές υπογράμμισαν τη σημασία της ε, ενεργής συμμετοχής των πολιτών πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών κοινοβουλίων και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται για αυτή τη συνέλευση. Επίσης, οι βουλευτές είπαν πως είναι απαραίτητο να ενημερώνονται τόσο οι θεσμοί όσο και η πολιτική της Ένωσης έτσι ώστε η συνέλευση να είναι πιο δημοκρατική και αποδοτική και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Οι βουλευτές επίσης θύμισαν ότι όπως συμβαίνει και στα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές αναφέρθηκαν στο ρόλο του Συμβουλίου ως άνω βουλής και τη διάκριση των εξουσιών επί τη βάση του άρθρου 4 της συνθήκης για τη χρήση της πλειοψηφίας και της απλής νομοθετικής διαδικασίας και τα ε, μιλήσαμε και για τα πολιτικά θέματα και το Μητρό της Διαφάνειας και το άρθρο 50 ως θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην συνέλευση. Αυτά όλα τα θέματα δεν είναι αρμοδιότητα της ε, υποψήφιας αντιπροέδρου. Οι βουλευτές αναφέρθηκαν επίσης στην ανάγκη να εξεταστούν μεταρρυθμίσεις για τα, τη κλιματική αλλαγή, τη διακυβέρνηση, την οικονομική και τις κοινωνικές πολιτικές. Τέλος, οι βουλευτές θεωρούν ότι η τα απορίσματα αυτής της συνέλευσης που θα μπορούσαν να οδηγήσει στην έναρξη της ε, ε τροποποίησης των συνθηκών θα ε, είναι τεραστία σημασία. Άρα λοιπόν όπως εμβαθύνατε στις γραπτές σας απαντήσεις για το θέμα της ε, συνέλευσης θα μπορούσατε ίσως στην ε, αρχική σας εισήγηση να τονίσετε, να στηρίξετε τις προσπάθειες του Ευρωκοινοβουλίου που στόχο έχουν να έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας, δικαίωμα έρευνας και άρα να παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης. Εγώ θα ε, παρουσιάσω στους συναδέλφους και στους συναντονιστές των ομάδων ε, μια σχετική επιστολή που θα υποβάλουμε στον πρόεδρο σας όλοι ώστε όντως να αναλάβουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω στις παρατηρήσεις σας να αναφερθείτε στη νέα στρατηγική και τα δικαιώματα των ανηλίκων. Ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλές στην Εύα Κόπατς, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, συντονίστρια του Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των ανηλίκων. Η Κομισιόν θα ε, πρέπει να μας πει πώς σκοπεύει να εφαρμόσει τέτοιες στρατηγικές και πώς θα αντιμετωπίσει προβλήματα όπως η εκμετάλλευση της φτώχειας των παιδιών και άλλα. Επειδή είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα, θα δώσω αμέσω το λόγο στην κυρία Ντουμπράφκα Σουίτσα. Ε, έχετε 15 λεπτά για την εναρκτήριά σας ομιλία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτή, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερω που βρίσκομαι εδώ και ω συνάδελφο και ω υποψήφια αντιπρόεδρο ε, για τη δημοκρατία και τη δημογραφία. Το... Νιώθω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σα στο σπίτι μου. Πριν από έξι χρόνια εξελέγει μέλο ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη κρατική αντιπροσωπεία μετά την προσχώρηση τη Κροατία το 2013 και με ιδιαίτερη χαρά ε, και τιμή επανεξελέγην ε, και για δύο συνεχείς χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη κοινοβουλευτική θητεία. Αυτή είναι η τρίτη μου δηλαδή κοινοβουλευτική θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο που βρίσκομαι εδώ σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα που θα ήθελα να μου δώσετε την εμπιστοσύνη σας για ένα χαρτοφυλάκιο που έχουμε συζητήσει επανειλημμένο στα τελευταία έξι χρόνια σε πολλέ συζητήσει που είχαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρωθήκαμε στα έξι. Πώ ε, να δώσουμε περισσότερο λόγο στους Ευρωπαίους πολίτες για το μέλλον και να μπορέσουν να το διαμορφώσουν και αυτοί. πώ θα δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη σε όσου νιώθουν ε, αλωτριωμένοι και αποδεσμευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ε, θα τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν όλες αυτές τις ρηξιγέλευθες αλλαγές και τις μεταβάσεις που χρειάζονται. Ε, ήμουν και εκπρόσωπος ε, του τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ήμουν δήμαρχος στο Ντούμπροβνικ ε, και μέλος της κρατικής αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδα λοιπόν ε, από πρώτο χέρι μερικές αρνητικές σκέψεις και απογοητεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών που νιώθουν ότι έχουν χάσει τον έλεγχο της ζωής τους. δεν νιώθουν ότι δεν έχουν κανένα λόγο σε διαμόρφωση ε, της, του μέλλοντός τους και ο τρόπος διαβίωσης τους, η σταδιοδρομία τους, όλα αυτά εξελίσσονται με ταχύτερο αριθμό που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Έτσι χάνουν την εμπιστοσύνη τους ε, στα θεσμικά όργανα που κανονικά έχουν σκοπό να τους εξυπηρετούν και να τους ε, να μεριμνούν για αυτούς. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και να δούμε ε, τους γενεσιουργούς λόγους αυτής της αποστασιοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών. Και δεν είναι τόσο το θέμα του, του δημοκρατικού έλλειμματος, αλλά του δημογραφικού έλλειμματος. Τα επόμενα χρόνια θα μιλήσουμε εκτενώς ε, για την κλιματική και την ψηφιακή μετάβαση. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να μιλούμε όλο και περισσότερο για μία από τις βαθύτερες αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η δημογραφική αλλαγή. Είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει εκατομμύρια Ευρωπαίους και φαίνεται σε πολλές γωνιές της Ευρώπης. Συνεπιφέρει και πολλές προκλήσεις αλλά και πολλές ευκαιρίες. Οι δημογραφικές αλλαγές θα ε, διαμορφώσουν το τοπίο των πολιτικών, της δημοκρατίας και των κοινοτήτων μας. Όσοι μείνουν πίσω από την πρόοδο, από την πρόοδο και τη μετάβαση, είναι αυτοί που θα νιώσουν περισσότερο και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη φωνή στους Ευρωπαίους, την ευκαιρία να ξανακατακτήσουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την κοινότητά τους, ε, τη ζωή τους, την κοινωνία στην οποία διαβιούν. Γι' αυτό και είμαι ένθερμη υπέρμαχος της ιδέας της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Η πρόταση αυτή υπευλήθη από την σαν πρόεδρο Φόντερ Λάιεν και χαίρομαι που θα πρωτοστατήσω στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οργάνωση της διάσκεψης. Εκεί θα συμμετέχουν πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως νέοι, αλλά και μέλη της κοινωνίας των πολιτών και εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων. Και όλοι αυτοί θα συμμετέχουν ισότιμα, επίσης όρις. Θέλουμε ξεκάθαρους στόχους, διαφανή συζήτηση και μία επακολούθηση, μία συνέχεια σε αυτά που θα συμφωνηθούν. Και μάλιστα αυτό το έχουμε συζητήσει εκτενώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δει στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Υπάρχει και η βούληση τώρα, αλλά και η κατάλληλη δυναμική να συνεργαστούμε για να στεφτεί με επιτυχία αυτή η πρωτοβουλία. Και τίποτα δεν δείχνει καλύτερα αυτή την ανάγκη από το ρεκόρ προσέλευση τη κάλπη στι τελευταίε ευρωεκλογέ. Πάνω από το 50% των Ευρωπαίων πολιτών ψήφισαν. Θέλουν να έχουν λόγο και αυτοί. Δείχνει την λαχτάρα του για και τη διάθεσή τους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία δεν είναι μόνο ψηφίζουμε μια φορά κάθε πέντε χρόνια. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θέλει να καταστήσει την ε, Ευρωπαϊκή Δημοκρατία μια ζωντανή έννοια που ξεπερνά την ε, εποχή των ε, ευρωεκλογών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού θα εστιαστούμε και πόσο φιλόδοξοι θα πρέπει να είμαστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η σαν πρόεδρος ε, έθεσε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα αναγγέλλοντα την έναρξη της διάσκεψης ε, το 2020 και διετή διάρκεια. Οπότε, αν μου δώσετε την έγκρισή σας, θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο και όλους τους άλλους ενεχομένου για να συμφωνήσουμε στην έννοια, τη δομή, τον τύπο, το χρονισμό, το χρονοδιάγραμμα και την εμβέλεια της διάσκεψης. Θα προτείνω σε έγκαιρο, σε πρώιμο στάδιο της ε, ανάληψης των καθηκόντων μου, της ιδέας μου και προσβλέπω σε συνεργασία και διάλογο μαζί σας γιατί εσείς εκπροσωπείτε τους ψηφοφόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι αν συνεργαστούμε θα φέρουμε σε αίσιο πέρα στη διάσκεψη, γιατί αυτό είναι ο σκοπό μα. Δεν θα έρθω τώρα σε λεπτομέρειε στη συζήτησή μα. Θα σα ε, αναφέρω ενδεικτικά δύο-τρει αρχέ που θα πρέπει να ε, είναι τα θεμέλια της διαδικασίας. Πρώτη ιδέα, πρώτη αρχή. Θα πρέπει να φτάσουμε σε όλους τους Ευρωπαίους. Στόχος μου είναι να με ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν λόγο για τον τρόπο διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για τα αποτελέσματά της. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους Ευρωπαίους παντού στην Ευρώπη, να αφουγκραστούμε τις ελπίδες, τις προσδοκίες τους, τις ανησυχίες τους που ε, συνδέονται φυσικά με τη ζωή τους με την καθημερινότητά τους. Αφορούν το κλίμα, το, την οικονομία, την ψηφιακή ανάπτυξη, τη παγκόσμια, τις παγκόσμιες αλλαγές και τις δημογραφικές αλλαγές. Η σαν πρόεδρος μου ζήτησε να βρω τρόπο για να εξασφαλίσω ευρύτατη συμμετοχή, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω του διαδικτύου και να γίνει εύκολη πρόσβαση στη διάσκεψη. Αυτή θα είναι η κορυφαία μου προτεραιότητα. Πρώτη ιδέα. Ιδέα δεύτερη. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να μονοποληθεί από ένα κόμμα, έναν άνθρωπο ή ένα θεσμικό όργανο, ούτε από ένα τμήμα της Ευρώπης. Θα πρέπει να είναι μια συλλογική ομαδική προσπάθεια. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερως και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεργαστώ στενά με τον Αντιπρόεδρο για τις διοργανικές σχέσεις και τις προβλέψεις και τον Αντιπρόεδρο για, τις, για τη διαφάνεια και τις αξίες. Θα φροντίσουμε ώστε να στεφτεί με επιτυχία αυτή η πρωτοβουλία που θα είναι σημαντικό ιδιαίτερα στην πρώτη φάση και θα πρέπει να βρούμε κοινό έδαφος για να δούμε πώς θα προωθήσουμε το σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων, το speech and candidate και την ιδέα των υπερεθνικών ψηφοδελτίων. Αυτό θα απασχολεί στο πρώτο τμήμα τη θητείας μα. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Αντιπρόεδρος Γιώροβα θα ηγηθεί αυτού αυτή τη συζήτηση, αλλά θα συνεργαστούμε μαζί τη για όλε τι πτυχέ τη διάσκεψη. Η ενίσχυση τη δημοκρατία τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει χωρί ενεργό συμμετοχή, χωρί. Η ενίσχυση της δημοκρατίας δεν νοείται χωρί το πιο σημαντικό φορέα, το πιο σημαντικό θεσμικό όργανο που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει ε, εκπροσωπεί την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Και θα συνεργαστώ και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο σε όλα τα στάδια της διάσκεψης. Και η τρίτη μου ιδέα είναι ότι η διάσκεψη αυτή θα πρέπει να αποφέρει καρπούς, να έχει αποτελέσματα. Γιατί καλός ο διάλογος, αλλά δεν είναι αυτός Χρειάζεται κατανόηση ε, και φυσικά ανάληψη δράσης και ό,τι συμφωνηθεί θα πρέπει να εφαρμοστεί, να περάσουμε από τα λόγια και στα έργα. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί πολλές φορές συμφωνούμε, αλλά δεν εφαρμόζουμε πάντα τα συμφωνηθέντα. Είναι ε, ρητή δέσμευση της εκλεγής σας Προέδρου στις πολιτικές της κατευθύνσεις και θα συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με τους συναδέλφους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες τις ε, επιτροπές, εδώ είστε παρό, παρούσες πέντε επιτροπές, αλλά θα συνεργαστώ με όλες τις επιτροπές και όλα τα θεσμικά όργανα για να εφαρμόσουμε τα συμφωνηθέντα. Μία ουσιαστική και επιτυχής διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα είναι σημαντικό εργαλείο για την, για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και συμμετοχή στη δημοκρατία μας. Όπως είπε και προηγουμένως, το κλειδί της ενδυνάμωσης της δημοκρατίας μας έγκυται στην ε, παρουσίαση και ε, αντίληψη του λόγου της. Νομίζω ότι ένα από τα σημεία που δεν ε, επεξεργαστήκαμε αρκετά είναι το θέμα των δημογραφικών αλλαγών. Αυτό το ξέρουν πολλές χώρες, γιατί είχαμε παρατεταμένες περιόδους μείωσης του πληθυσμού που επηρεάζουν ε, ολόκληρη τη χώρα. Για κάποιες περιοχές της Ευρώπης ε, αυτό το θέμα φαίνεται αφηρημένο ή άσχετο, αλλά για άλλε ε, περιφέρειες και μάλιστα για πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και για αγροτικές περιοχές ολόκληρη την Ευρώπη, το θέμα αυτό είναι πολύ απτό και ανησυχεί τον κόσμο. Τον κόσμο που εξαρτάται από τοπικές υπηρεσίες και βλέπει ταχυδρομεία, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία να κλείνουν ή ε, οι περαστικές γραμμές να μειώνονται. Αυτή είναι η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές, οπότε οι δημογραφικές αλλαγές είναι μια απτή και σημαντική ανησυχία που βλέπουν τα παιδιά τους να μην έχουν ευκαιρία για δουλειά ε, ή για σπουδές. Και αυτό ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερω όσου μεγαλώνουν τα παιδιά του ε, σε δύσκολε συνθήκε και προσπαθούν να συμφιλειώσουν την προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Φυσικά το προσδόκιμο ζωής ε, έχει μεγαλώσει και η υγεία μας έχει βελτιωθεί. Αλλά το γεγονός αυτό συνδυάζεται με άλλες προκλήσεις, είτε οικονομικές, το συνταξιοδοτικό θέμα, το ζήτημα και του κοινωνικού ιστού και το, τα ζητήματα της υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την κατανόησή μας για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό και πρόκειται να γίνει μια εκτεταμένη χαρτογράφηση της κατάστασης για να δούμε πού βρίσκονται τα προβλήματα και πώς να βοηθήσουμε κυρίως στις περιοχές που το χρειάζονται. Να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις και να προσελκύσουμε επενδύσεις. Αν μου δώσετε την έγκρισή σας, εσείς, οι ευρωβουλευτές, θα εξετάσω όλες τις πτυχές των δημογραφικών αλλαγών και το πώς επηρεάζουν τις διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε. Πρώτον, ε, θέλω να κοιτάξουμε το θέμα της γύρανσης που είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην κοινωνία μας. Αυτό αφορά ε, τα συνταξιωτικά συστήματα, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και τον εργασιακό μας βίο. Συνοδεύεται και από πολλές ευκαιρίες. Θα πρέπει να υπάρχει η μεταβίβαση της γνώσης από γενιά σε γενιά και οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι να είναι και δραστήριοι και ενεργοί πολίτες. Θα προωθήσω μια πράσινη βίβλο για τη γύρανση, για να εκτιμήσουμε τι χρειάζεται να γίνει και τι μπορεί να γίνει, ιδιαίτερα για να βοηθήσουμε την ενεργό γύρανση και να προετοιμάσουμε τα στήματα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα γίνει σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο σας και φυσικά με τα κράτη-μέλη που έχουν τις αρμοδιότητες στους περισσότερους από αυτούς τους τομείς. Δεύτερον, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στις υπαίθριες περιφέρειες που πλήττονται σφοδρότατα από την ε, αποψήλωση του πληθυσμού, την αστιφιλία, τη διαρροή εγκεφάλων, τη μείωση των υπηρεσιών και τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Επίσης θα συντονίσω ε, ένα όραμα μακροπρόθεσμο ε, στη συνεργασία με τους ΟΤΑ και τις περιφερειακές αρχές για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές τους ε, και να ακούμε και τα θέματα που τα γνωρίζουν είναι καλύτερα. Θα σταθώ στη διαρροή εγκεφάλων για να υποστηρίξουμε τις πιο ε, ευάλωτες περιφέρειες και με την εγγύηση για την νεολαία. Τρίτον, και ως εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα συντονίσω την εργασία ε, για να συμφιλιώνεται καλύτερα ο εργασιακός με τον ιδιωτικό βίο και οικογενειακό. Και τελευταίο, χωρίς αυτό να είναι και το λιγότερο σημαντικό και έτσι έρχομαι να απαντήσω στην ερώτησή σας αξιότιμε πρόεδρε και θα επεκταθώ στη συνέχεια. Με ρωτήσατε για τα παιδιά. Βεβαίω, θα πρέπει να επενδύσουμε στου ανηλίκου και θα πρωτοστατήσω σε αυτό. Άλλωστε, ήταν και προτεραιότητά μου καθ' όλη τη σταδιοδρομία μου στην πολιτική. Δεν υπάρχει πολυτιμότερη επένδυση από την επένδυση στα παιδιά μα. Αν μπορούμε να την ονομάσουμε επένδυση. Ε, θα συντονίσω τις εργασίες για μια νέα εγγύηση για τα παιδιά και θα παρουσιάσω και μια σύμβαση για τα δικαιώματά τους. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εκτενώς. Ε, χαίρομαι για όλες τις ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάτι προσωπικό. Ε, έζησα τη χώρα μου να ανακτά την ε, ανεξαρτησία της, τον εκδημοκρατισμό της και τη μετάβαση. Και με μεγάλη λοέστημα ε, ευθύνης αλλά και ταπεινότητας αποδέχτηκα αυτή την αποστολή με την οποία με επιφόρτησαν για να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις στις αλλαγές που μας επηρεάζουν όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όλα γίνονται χάρη στις θυσίε εκείνων που προηγήθηκαν για να οικοδομήσουμε όλοι μαζί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν με εγκρίνετε, ε, είμαι αποφασισμένη και θα έχω και τη μεγάλη τιμή σε συνεργασία μαζί σας να προωθήσουμε όλα αυτά τα θέματα την επόμενη πεντέτεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω τις ερωτήσεις σας με ανυπομονησία. Ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε που επαναλάβατε τη δέσμευση σας που για μας είναι πολύ σημαντική για τη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης και επειδή επίσης ε, μιλήσατε για το σημαντικό ρόλο που θα έχει σε αυτήν το κοινοβούλιο μας. Δεν μπορεί να είναι ένα ε, ρόλος παρατηρητή αλλά πρωταγωνιστικός ρόλος. Αρχίζουμε με τον πρώτο γύρο των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Ε, πρώτη ερώτηση από την κυρία Ντανούτα Χουμπνέρ, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Έχετε το λόγο. Κυρία Αντιπρόεδρε, υποψήφια Αντιπρόεδρε, ε, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για την περιστατωμένη σα εισήγηση ε, για την σημερινή συζήτηση. Εσύ, εμεί εδώ είμαστε συνάδελφοι από διάφορε επιτροπέ τη Ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όμως η Βασική Επιτροπή είναι η Επιτροπή των Συνταγματικών Υποθέσεων που τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, ασχολείται με το προβληματισμό για το μέλλον της Ευρώπης ε, ως θέμα προτεραιότητας και νομίζω πως θα παραμείνει και θα μας, συνεχίσει να μας απασχολεί αυτό το θέμα. Γι' αυτό και η μελλοντική σας εργασία θα είναι πολύ σημαντική για μας αυτή την εδώ την Επιτροπή. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν πώς βλέπετε εσείς τη συνεργασία με τους μεμονωμένους ευρωβουλευτές αλλά και με το Ευρωκοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο και την Επιτροπή μας. Ε, πώς βλέπετε λοιπόν εσείς τη συμμετοχή σας σε όλα τα στάδια αυτής της πολιτικής διαδικασίας προπαρασκευής αυτού του κύριου project μας που θα ξεκινήσει αμέσως ε, με τη θητεία σας. Γιατί πιστεύω πως η διαδικασία προπαρασκευής αυτής της συζήτησης και αυτής της συνέλευσης μπορεί η ίδια αυτή η προετοιμασία να έχει μεγάλη αξία ε, για την ε, διοργάνωση αλλά και για την υλοποίηση της συνέλευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σας ευχαριστώ που την ε, θέσατε εξ αρχής, γιατί όπως είδατε και από την εισαγωγική μου ε, ομιλία, ε, η συνέλευση θα είναι ένα κύριο κομμάτι του χαρτοφυλακίου μου. Προσπαθώ να παρακολουθώ τι κάνετε εδώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, αλλά και μέσα από τις Ολομέλες παρακολουθούσα τις εκθέσεις του κυρίου Μπροκ, της κυρίας Μπέ, αφαιρέσω έπειτα την έκθεση του κυρίου Φερχόφστατ και την τελευταία επίσης. Και έχω λοιπόν παρακολουθήσει τι κάνετε σε αυτό το τομέα. Χωρίς εσάς, χωρίς το ε, κοινοβούλιο, εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω την συνέλευση αυτή. Έρχομαι λοιπόν στην επιτροπή σας και θα συμφωνήσουμε για το ε, ε, πεδίο, για το εύρος, για το χρονοδιάγραμμα, για τα θέματα νομίζω θα πρέπει να μείνουμε και να μείνουμε σε αυτούς τους έξι πυλώνες που ε, περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της υποψήφιας Πρόεδρου, δηλαδή ε, το νέο το σύμφωνο για το κλίμα, ψηφιακή ε, ε, οικονομία, οικονομία για τους λαούς, ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και μια νέα όθεση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Νομίζω πως αυτό θα πρέπει να είναι το πεδίο των συζητήσεων της συνέλευσης και θα είναι το πρώτο μου έργο εντό των πρώτων 100 ημερών. Θα έρθω λοιπόν εδώ και θα δούμε από κοινού πώς θα προχωρήσουμε. Είμαι βεβαία ότι θα πρέπει όλα αυτά να προετοιμαστούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο βέβαια, αλλά εσείς θα είστε νομίζω οι πρώτοι που θα, ε, ε, με τους οποίους θα έρθω σε επαφή. Κυρία Χούμπνερ, ναι, συμπληρωματική ερώτηση σύντομα. Είδα στο βιογραφικό σας ότι παραδοσιακά ήσασταν, ήσασταν τοπική πολιτικός και αυτό το εκτιμώ πολύ. Ως ε, ε, ε, ε Πώς βλέπετε τη συμμετοχή των πολιτών στην συζήτηση ε, ώστε να μπορέσουν μετά να ιδιοποιηθούν τη συμφωνία και τα πορίσματα, τα αποτελέσματα αυτής της συνέλευσης. Κοιτάξτε, Δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία χωρίς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Όπως είπα στην εισήγησή μου, έχω υπηρετήσει σε διάφορα επίπεδα της αυτοδιοίκησης, χωρίς, όπως σας είπα, αυτήν την συμμετοχή της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα πράγματα αγαστά. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν η ΜΚΟ, η κοινωνία των πολιτών, η αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό είναι ευκολότερος τρόπος για να φτάσουμε στους πολίτες, ως όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για το κοινό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση από το συντονιστή της Σοσιαλιστικής και Δημοκρατής Ομάδας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Δόμενα Ιστεβες. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία ε, Σούιτσα, υποψήφια αντιπρόεδρα ο κύριο Εμεί, οι σοσιαλιστέ και δημοκράτε, πιστεύουμε ότι η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για να ε, ξαναδούμε τι ε, συνταγματικέ μεταρρυθμίσει και τι θεσμικέ που χρειαζόμαστε τα επόμενα χρόνια. Για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει νέε πολιτικέ όπω αυτέ που αναφέρατε απέναντι στι μεγάλε διεθνεί προκλήσει και να παίρνει αποφάσεις πιο δημοκρατικά και πιο γρήγορα. Η εκλεγμένη πρόεδρος ε, δήλωσε ότι προτίθεται να δώσει συνέχεια στις συμφωνίες αυτής της ε, διάσκεψης και μεταξύ αυτών και νομοθετική και ε, μεταρρύθμιση των συνθήκων. Ταυτόχρονα όμως η κυρία Φόντερ Λάιεν έχει ένα πρόγραμμα πολιτικό σε έξι γραμμέ, νέο πράσινο deal, εμβάθυνση τη ΟΝΕ, κοινωνικό πυλώνα, ασφάλεια, μετανάστευση, εξωτερική πολιτική και νέα όθηση στη δημοκρατία. Κατά την άποψή μα, αν δεν υπάρξουν νομοθετικέ πρόοδοι ή αναθεώρηση των συνθήκων, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί αυτό το πολιτικό πρόγραμμα που είναι και δικό σα. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή, τι συμμερίζεστε, γιατί στι γραπτέ σα απαντήσει στη σελίδα 6, αναφερόμενοι στην ενδεχόμενη η αναθεώρηση των συνθήκων προσθέσατε ότι αυτό θα γίνει σε περίπτωση που θα χρειαστεί. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πώς μπορεί να διαπιστώσετε ακολουθώ τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της εκλεγμένης Πρόεδρου και φυσικά αυτό θα ε, είναι ένα ενδεχόμενο. Αλλά Ας πάμε πρώτα στην Ήπεθρο, ε, ας πάμε πρώτα στα βουνά, στα μακρισμένα μέρη και στις πρωτεύουσε και να συζητήσουμε με τους πολίτες. Και μετά από μια διετία, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το διάστημα χρειάζεται, θα δούμε τι θα έχουν πει οι πολίτες. Need Αν χρειάζεται αλλαγή, ε, τροποποίηση των συνθήκων, ε, εγώ είμαι πρόθυμη να το συζητήσω και όχι μόνο εγώ και όλοι σας είδα ότι ήταν ιδέα της Επιτροπής σας και είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο να είναι πιο ισχυρό και να έχει και περισσότερες εξουσίες. Και εγώ ευρωβουλευτής είμαι στο κάτω-κάτω. Υπέρ θα ε, ε, ταχθώ. Αλλά ξέρετε ότι είναι συλλογικό σώμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάζεται ομαδικά. Και αν είναι ομόφωνη ε, η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά, εγώ είμαι υπέρ. Υπάρχει αυτή η συνθήκη και αρκεί αυτή η συνθήκη να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που μας παρέχει. Ιδάλλως θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε για την τροποποίηση της συνθήκης. Ε, συμπληρωματική ερώτηση του κυρίου Ρουίς Δεβέσα. Ευχαριστώ πολύ. Εν πάση περιπτώσει, σας θυμίζω ότι το κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες ήδη έχει εγκρίνει τρεις εκθέσεις αρκετά σημαντικές για τις προόδους στην ολοκλήρωση εντός της συνθήκης. Έκθεση Μπροκ Μπρέσο ή Μπρέσο Μπροκ. Και κατά κάποιο τρόπο επίσης έκθεση της κυρίας Περβάνς Μπερές. Και μετά έχουμε την έκθεση Φερχόφστατ και Χάουραγγι για πιο προχωρημένες ε, μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια των συνθήκων. Συμφωνείτε με τις εκθέσεις αυτές. Την προσωπική σας άποψη ρωτώ. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να διαβουλευτείτε με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης. Παρακαλώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Φυσικά και τις γνωρίζω τις εκθέσεις αυτές και τις υπερψήφισα στην Ολομέλεια Έλαβα και το λόγο μάλιστα στι συζητήσεις. Και ασθενίζομαι το περιεχόμενό τους. Αλλά, ε, όπως σας είπα, βήμα-βήμα θα προχωρήσουμε. Και είδομεν. Έχουμε αρκετό χρόνο για να αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Συμφωνώ πάντως, γιατί πιστεύω ότι το κοινοβούλιο είστε, είμαστε άμεσα εκπλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και έχει το κυριότερο και το μεγαλύτερο λόγο μεταξύ όλων των άλλων οργάνων το Κοινοβούλιο σχετικά. Ας συνεργαστούμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή και θα συνεχιστεί η συζήτηση. Φυσικά είμαι υπέρ. Ναι, ναι. Ε, είχατε υπερψηφίσει την έκθεση. Είστε υπέρ. Είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε. Η επόμενη ερώτηση θα γίνει από τον κύριο Πασκάλ Ντουιρόν, που είναι ο συντονιστής της ομάδας Renew Europe. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που μου δώσετε και το λόγο στα γαλλικά. Κυρία υποψήφια αντιπρόεδρε, μας εξηγήσατε ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δώσουμε νέα δυναμική στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, να την αναζωογονήσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα με τους Ευρωπαίους πολίτες. Και είπατε το Νοέμβριο θα καταθέσετε και σχετικές προτάσεις. Ίσως όμως καλό θα ήταν να αλλάξει η μεθοδολογία. Αντί να υποβάλλετε τις προτάσεις τον Νοέμβριο, να ακούσετε τις δικές μας προτάσεις. Όταν θα αναλάβετε τα καθήκοντά σας, να λάβετε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής μας για τη διάσκεψη της Ευρώπης. Γιατί και εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών έχουμε δικαίωμα να έχουμε και προτάσεις και ιδέες και να τις ε, υποβάλλουμε και το ίδιο και το, το Συμβούλιο. Είπατε ότι θέλετε να εμπλέξετε τους πολίτες. Μα πάνε χρόνια που αναμειγνύουμε τους πολίτες με την πρωτοβουλία των πολιτών και ούτω καθεξής. Θα μπορούσατε να διανεθείτε το εξή. Ή να επιτρέψουμε στους Ευρωπαίους πολίτες να ψηφίζουν και να αποφασίζουν και όχι μόνο να λένε τη γνώμη τους και να τους αφογκράζονται οι θύνοντες πολιτικής και μετά να λαμβάνουν τις αποφάσεις στο όνομά τους. Οπότε, αν υπήρχε ένα κολέγιο, ένα συλλογικό όργανο ε, ε, Ευρωπαίων πολιτών σε αυτή τη διάσκεψη Ευρώπης να έχει την ίδια δύναμη για λήψη απόφασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πασκάλ Τουιχό. Καταρχήν, να σας πω χρόνια πολλά, γιατί έχετε και γενέθλια. And then, and then let's be... και φυσικά να είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς. Γνωρίζουμε ότι δεν αρχίζουμε από το μηδέν. Ήδη είχαμε και πρωτοβουλίες και μέσα και εργαλεία διάφορα. Θυμάς, ε, φανταστείτε, είχαμε 1.800 διαλόγους πολιτών με τη συμμετοχή 200.000 Ευρωπαίων πολιτών που πήραν μέρος αυτούς τους 1.800 διαλόγους σε 635 περιοχές έγιναν, σε 635 μέρη. Είχαμε ήδη δηλαδή διάλογο με τους πολίτες, απλώς θα πρέπει να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας. Εσείς με ρωτήσατε για τους πολίτες. Έχουμε και την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Και εκεί είχαμε τέσσερις επιτυχημένες πρωτοβουλίες των πολιτών. Το δικαίωμα στο νερό, ε, η απαγόρευση της γλυφοσάτης, Έχουμε δηλαδή μέσα και μηχανισμούς, απλώς θα πρέπει να τα μεγιστοποιήσουμε, να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας. Και φαίνεται να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της άμεσης δημοκρατίας και των εκπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών, αν υπάρχει μια σύγκρουση, αλλά όχι. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ήδη μια πολύ καλή πρωτοβουλία για να αφογκραστούμε τους πολίτες και μπορούμε να τις διευρύνουμε. Και από τη στιγμή που οι μισοί Ευρωπαίοι έλαβαν μέρο σε εκλογέ, δηλαδή αυξήθηκε κατά πολύ το ποσοστό προσέλευση στι κάλπε σε σχέση με τι προηγούμενε ευρωεκλογέ. Αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πηγαίνουμε επί τόπου, μιλούμε στου πολίτε, αφού τι ανησυχίε του, τι προσδοκίε του. Και φυσικά θα ακούσω και τις δικές σας προτάσεις πρώτα. Και βλέπω ότι ο χρόνος μου πέρασε. Θα απαντήσω στη συνέχεια. Χρόνια πολλά και από μένα. Δεν έχετε το λόγο για περώτηση. Ναι, συνεχίζω, γιατί κυρία Αντιπρόεδρε, αναφερθήκατε και στη γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. <laughs> Απόδειξε τα γενέθλιά μου και σας ευχαριστώ που το επισημάνατε. Τώρα πιο σοβαρά. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο δημογραφικό ζήτημα από μία όμως πιο πολιτική σκοπιά. Μιλήσατε για τη γύραση του πληθυσμού και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή πνέουν πολύ αρνητικοί άνεμοι στην Ευρώπη. Και κυκλοφορεί μία θεωρία που επισημαίνει τον κίνδυνο της μεγάλης αντικατάστασης του ευρωπαϊκού πληθυσμού εμ, χριστιανικών καταβολών με τις γνωστές ιστορικές μας αξίες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, γιατί είμαστε ακριβώς στο επίκεντρο του χαρτοφυλακίου σας, γιατί είναι η δημογραφία, του χαρτοφυλακίου σας, τι γνώμη έχετε για αυτή τη θεωρία και πώς βλέπετε αυτό το πιθανό κίνδυνο της αντικατάστασης ε, των μέχρι τώρα γνωστών σε εμά ευρωπαϊκών αξιών. Άμα επιτρέπετε, θα σας πω ευθέως ότι δεν πιστεύω στη θεωρία αυτή. Πάντως, είναι αλήθεια ότι ζούμε έξι χρόνια περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Το προσδόκιμο ζωής μας έχει αυξηθεί κατά έξι χρόνια. Οπότε η γύρανση είναι κάτι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να το φροντίσουμε. Αλλά αυτό θα το, θα το συζητήσουμε αργότερα. Πάντως, και το ποσοστό γεννητικότητας μειώνεται, αλλά υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης, της νόμιμης μετανάστευσης, με την οποία δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί χωρίς νόμους μετανάστες, η αγορά εργασίας μας το 2070, αν συνεχίσει ο ρυθμός αυτός, θα χάσει 25% του εργατικού δυναμικού της. Οπότε χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ένα μακροπρόθεσμο όραμα και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και γι' αυτό ε, το χαρτοφυλάκιο της δημοκρατίας με τη δημογραφία είναι σημαντικό, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, συνυφασμένες οι δύο έννοιες της δημοκρατίας και της δημογραφίας. Αλλά θα το εξηγήσω πιο διεξοδικά αργότερα, γιατί ο χρόνος μου πέρασε. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντάμιαν Μπουσελάκερ από τους πράσινους. Όπως είπατε, οι τελευταίες ευρωεκλογέ είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή τη τελευταία 20 ετίας, με πολλή υποστήριξη για τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, κυρίως από τους νέους που μας ζητούν μια πραγματική αλλαγή θα κάνετε μια διάσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να σας ξαναρωτήσω για τις λεπτομέρειες. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα συμμετέχουν ε, ουσιαστικά οι πολίτες και οι εθνικοί βουλευτές και πώς δεν θα επαναλάβετε τα λάθη του παρελθόντος και επίσης ποιες είναι οι συγκεκριμένες ε, συνέπειες και τα αποτελέσματα θα βγάλετε, τα συμπεράσματα. Δηλαδή αν χρειαστεί θα τροποποιήσετε και τις συνθήκες όπως ρώτησαν και άλλοι συνάδελφοι προηγουμένω. Όπως σας είπα, ήρθα εδώ να σας μιλήσω. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς ε, θα συνδιαλλαγούμε με τους πολίτες. Ε, κάποιος με ρώτησε ε, και ποιος θα τους διαλέξει τους πολίτες. Στα δημαρχία οι Φιλανδοί τώρα βγάζουν στις δημόσιες βιβλιοθήκες όλο το νομοθετικό πρόγραμμα, τα νομοσχέδια αυτό μπορεί να θεωρείται πιο συντηρητική προσέγγιση ή μπορεί να γίνουν περιοδίες όπως κάνει ο πρόεδρος Μακρό από πόλη σε πόλη στη Γαλλία ή μπορεί να γίνει επιγραμμική διαβούλευση. Θα είναι ε, απολύτως ε, ανοιχτά όλα αυτά, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς. Θα ε, συζητήσουμε με τους πολίτες, θα τους ρωτήσουμε και θα συμφωνήσουμε για τα αποτελέσματα. Αυτή ήταν η τρίτη μου ιδέα. Αν δεν έχουμε απτά αποτελέσματα αν δεν καταγράψουμε κάπου ε, ε, τι συζητήσαμε και τι συμφωνήσαμε και δεν δώσουμε συνέχεια, θα είναι κενό γράμμα όλα αυτά. Ας συνεργαστούμε λοιπόν και ας προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Φυσικά θα υπάρξει και ένα συμβούλιο, ένα συμβουλευτικό όργανο, στο οποίο θα προεδρεύω εγώ, αλλά θα συμπροεδρεύει κάποιος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι μια πρωτοβουλία ε, μονοπόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν θα έρθουμε για διαβούλευση όμως μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά θα πάμε και στους πολίτες. Γιατί αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν με τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογέ. Θέλουν οι πολίτες να έχουν λόγο να συνδιαμορφώνουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πράγμα που δεν ίσχυε πάντα στο παρελθόν. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Όπως είπατε, δεν αρκούν τα λόγια, πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα απτά έργα. Ε, ποιο, αυτό το συμβουλευτικό όργανο, η Επιτροπή αυτή, τι ρόλο θα έχει και θα μας υποστηρίξετε ε, στο να καταλήξει σε ουσιαστική συντακτική συνέλευση μετά ε, η διάσκεψη αυτή. ναι, κάποιο θα πρέπει να προεδρεύει ε, σε όλη αυτή την προσπάθεια, στη συμβουλευτική αυτή επιτροπή. Ε, είναι μια διάσκεψη, αλλά μια διάσκεψη που θα διαρκέσει δύο χρόνια. Ουσιαστικά είναι μικρές διασκέψεις παντού σε όλη την Ευρώπη. Αυτό έχουμε υπόψη. Βεβαίως, όποιο θέλει να συμμετέχει και έχει ιδέε. είναι ευπρόσδεκτος δεν θα πούμε εμείς δεν δεχόμαστε κάποιες ιδέες. Μην αμφιβάλλετε ότι θα δεχτούμε όλες τις ιδέες, ότι θα τις υποδεχτούμε μάλλον και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφεράσουμε σε ε, πολιτικές χειροπιαστές, γιατί μας στέλνουν μηνύματα οι πολίτες. The Επόμενη ερώτηση ο κύριος Άνεμανς, ε, συντονιστής της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία. Γεια σας κυρία Σούιτσα. Ζητώ συγγνώμη. Ε, ε, ε εξ ονόματος Επιτροπής ΑΦΚΟ. Σύμφωνα με την κυρία Φόντερ Λέιεν, έχει δημιουργηθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ε, ε, σε τι αποσκοπεί, ποιες είναι οι αρμοδιότητες ας πούμε του Έλληνα Επιτρόπου. Είναι μια συζήτηση που έχει αρχίσει τώρα με ε, τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και δεν έχει ξεκαθαριστεί, δεν έχει διευκρινιστεί. Υπάρχουν διάφορες αρμοδιότητες με βαβυλώνια γλώσσα, με μια κακοφωνία, με συγκεχημένες εντυπώσεις. Και ακόμα και η κυρία Φοντερ Λάιεν ε, χρησιμοποιεί αυτή τη σύγχυση ε, για να εκμεταλλευτεί ε, την κατάσταση και να θολώσει τα νερά γιατί η τριμερής που την έχει φέρει στην εξουσία έχει προβλήματα αυτό η συμμαχία. Και είδαμε πώς εξελέγει η πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι συνεννοήσεις είχαν γίνει με τις πέντε αστέρες. Ξαφνικά τώρα έχουμε επίτροπο για τη δημογραφία. Αλλά ε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ε, ε, έχουμε μια μαζική μετανάστευση η οποία, την οποία απορρίπτει στην τριπτική πλειονότητα των πολιτών αλλά δεν έχουμε χαρτοφυλάκιο για τη μετανάστευση και είναι και άγρια μετανάστευση ε, ανεξέλεγκτη που οργανώνεται καθημερινά. Οπότε, πώς ξαφνικά συνδέεται το δικό σας χαρτοφυλάκιο με τη μετανάστευση. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Έχετε δύο λεπτά. Τα πέρασα και όλα στα δύο λεπτά. Ένα λεπτό νόμιζα. Α, νόμιζα ότι είχα πέντε λεπτά. Καλά, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Έχω κι άλλη. Okay, Καλά, είμαι και ευέλικτο. Και πολύ ευέλικτο είστε, Πρόεδρε. Κύριε Άνεμαν, σα ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Καταρχάς, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ στα πολιτικά σα σχόλια για τι συμμαχίε για την κυρία ε, εκλεγμένη πρόεδρο Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Αλλά αν ενδιαφέρεστε για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ε, δυο ρόφους πιο κάτω γίνεται τώρα ακρόαση σχετικά. Δεν ξέρω τι συζητούν αυτή τη στιγμή, αλλά για τη δημογραφία και την δημοκρατία δεν θα έλεγα ότι είμαι θύμα εγώ αυτού του τίτλου του χαρτοφυλακίου σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο ε, και με εμπνέει. Και το είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία. Μίλησα για τη διαρροή εγκεφάλων. Μίλησα για τα προβλήματα που δυσαρεστούν τον κόσμο και εγκαταλείπει την, ύπεθ, εγκαταλείπει την ύπεθρο ε, τις χώρες ε, του κόσμου ε, και πηγαίνει από τις ε, περιοχές στην ε, πόλη. Αυτά είναι τα προβλήματα, αλλά η δημοκρατία και η δημογραφία είναι αλληλένδετες. Γιατί όσοι μένουν τα χωριά, εκεί που κλείνουν όπως σας είπα σχολεία, νοσοκομεία, ταχυδρομεία, ε, μειώνονται τα υπεραστικά δρομολόγια, για να μην πω καταργούνται τελείως. Τα είπα όλα αυτά εισαγωγικά. Εκεί ο κόσμος αρχίζει να κατηγορεί τη δημοκρατία για όλα αυτά που του συμβαίνουν. Και δεν πιστεύει πια στους δημοκρατικούς θεσμούς, σταματάει να ψηφίζει. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουν όλοι. Γι' αυτό διοργανώνουμε αυτή τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Θέλουμε να ακούσουμε όλους τους πολίτες. Και όχι μόνο μια φορά κάθε πέντε χρόνια στις ευρωεκλογέ σε καθημερινή βάση, επιγραμμικά ή εκτός διαδικτύου. Έτσι εξηγώ το χαρτοφυλάκιά μου για να δεν έχω χρόνο παραπάνω. Short, short Σύντομη συμπληρωματική ερώτηση. Θα είμαι σύντομος. Άκουσα μια φήμη. Ο κύριος Φερχόφστατ θα προεδρεύσει στη διάσκεψη αυτό. Ισχύει. είστε μέλος της Επιτροπής. Θα έρθω εγώ στην Επιτροπή σας και θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο ποιο θα στείλει συμπρόεδρο. Ε, αυτό είναι, υπερβαίνει τις δικές μου αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now, uh, Mr. Gert Bourgeois. Ο κύριος Χέρτ Μπουρζουά, συντονιστής ε, της ομάδας ECR. Ε, Ευχαριστώ. Ε, θέλω κύριε Πρόεδρε, να καλωσορίσω την υποψήφια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν είναι superstar. Ε, βασίζεται στην, ε, είναι ενωμένη στην πολυμορφία και βασίζεται στην επικουρικότητα. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την έκθεση Timmermans για την ενεργή επικουρικότητα. Σας ερωτώ, θα δώσετε συνέχεια στην έκθεση αυτή και πια. Και δεύτερον, κατά την άσκηση αυτή είστε πρόθυμοι να εργαστείτε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί υπάρχει προστιθέμενη αξία από τη συνεργασία. Αυτό θα έρθει ως αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα παραμείνει στα κράτη-μέλη με τις νομοθετικές τους αρμοδιότητες. Και μια τρίτη ερώτηση. Συμφωνείτε ε, ε, με το να θεσπιστεί η κόκκινη κάρτα όταν η πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων θεωρεί ότι μια νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν συνάδει με την επικουρικότητα. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουρζά. Ήταν πολύ α, ε, άμεσες ερωτήσεις, ιδιαίτερη τελευταία ευθύς ερωτήσεις μάλλον. Ε, σαφώς είμαι υπέρ της επικουρικότητας Μάλιστα κατοχυρώνεται στις συνθήκες μας και η επικορικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και είμαι αναφανδόν υπέρ. Και για τα μικρά θέματα τα κράτη-μέλη, για τα μεγάλα η Ευρώπη, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ. Για την τρομοκρατία, για τη μετανάστευση, για την ασφάλεια δεν μπορεί η χώρα μόνη της να αναλάβει τα θέματα, αλλά για την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισμό, μπορούν τα θέματα να διευθετηθούν σε, σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά και είμαι υπέρ της επικουρικότητας, φυσικά και θα τη διαφυλάξω. Και είμαι αρμόδια και για τον κοινωνικό πυλώνα. Φυσικά θα λάβω υπόψη τις εθνικές αρμοδιότητες, εννοείται, αλλά για τον κοινωνικό πυλώνα, εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί να μην το κάνουμε γιατί να μην βοηθήσουμε τον κόσμο ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη που οι χώρες υστερούν λίγο σε ανάπτυξη, σε ό,τι αφορά την κόκκινη κάρτα. Αρχικά έχουμε την κίτρινη κάρτα που χρησιμοποιήθηκε μέχρι στιγμής τρεις-τέσσερις φορές. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε την πράσινη κάρτα, έχουμε την κίτρινη, κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε και στην κόκκινη. Αλλά γιατί να μην τα συζητήσουμε όλα αυτά στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Και αν αυτό είναι το συμπέρασμα και το ζητούμενο, υπάρχει και κόκκινη κάρτα, γιατί όχι. Είμαι απολύτως διαλλακτική, ανοιχτή και συμμετοχική. Και αυτό είναι το πνεύμα που διέπει το νέο κολέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Μπουρζουά. Ευχαριστώ για την απάντησή σας προφανώς αυτά που αναφέρατε, τα παιδιά, την νεολαία, ε, την πολεοδομία, το σχεδιασμό, βεβαίως αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και είπατε ότι αυτά θα συζητηθούν στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Είστε πρόθυμοι να συζητήσετε εκεί και την αρχή της αναλογικότητας αρχή της απεικορικότητας αλλά και αρχή της αναλογικότητας ήδη περιλαμβάνονται. Ε, φυσικά και τις έχουμε κατά νου και τις λαμβάνουμε υπόψη. Και η αναλογικότητα είναι πολύ σημαντική αρχή. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε κανέναν επιπλέον. Ιδιαίτερα όχι τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Διατέλεσα δήμαρχος μίας σχετικά μικρής πόλης, αλλά γνωρίζω τι σημαίνει να εργάζεται κανείς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειάζονται λοιπόν αρμοδιότητες σε τέτοιο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και φυσικά και σεβασμό σε αρχή τη αναλογικότητα. Επικουρικότητα λοιπόν και αναλογικότητα ταυτόχρονα. The last speaker of the uh, είναι ο κύριος Σόλτς, εξ ονόματος της ομάδας της ΓΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρία υποψήφια Αντιπρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ήδη και από ό,τι φαίνεται η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης τώρα είναι μια πανάκια που βρήκαμε ε, για να εκδημοκρατήσουμε την πολιτική και ε, τις ε, συνθήκες στην κοινωνία. Η δημοκρατία όμως είναι πάντα κάτι το συγκεκριμένο και θα πρέπει να είναι και χωρίς αποκλεισμούς. Είπατε πολλά για την κατάσταση στην Ήπεθρο, έγινε μεγάλος λόγος για τις προκλήσεις ε, τις δημογραφικές στην κοινωνία. Τι γίνεται όμως αυτή τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Θέλω να σταθώ λίγο. Εσείς τι λέτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μας επιφυλάξετε τον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των στόχων, των ε, εργαλείων και των μέσων με συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών και σε συνεννόηση με το Συμβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρωτοστατήσει εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει από την αρχή να έχουμε αυτή την ε, προσέγγιση για το μέλλον της Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, με συμπερίληψη όλων. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς για την ερώτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ήδη έχω καλύψει ένα τμήμα τη απάντησης, αλλά όχι το σύνολο. Άπαντες θα συμπεριληφθούν στη διάσκεψη. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω θα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας πρώτα, να ακούμε ένα τον άλλον και να δούμε τι θα κάνουμε. Και τα εθνικά κοινοβούλια φυσικά θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό και είπα στον κύριο Μπουρζουά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς που έχουμε και όλα τα μέσα. Φυσικά και τα εθνικά κοινοβούλια θα είναι μέσα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τις προάλλες έλαβα μία επιστολή με 100 υπογραφές από 100 διαφορετικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και συνάντησα μερικέ από αυτές. Οπότε θα είναι παρούσες και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών. Φυσικά εννοείται να είστε βέβαιος ότι θα τους συμπεριλάβω όλους. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί θα συμπροεδρεύσουμε στη διάσκεψη αυτή. Οπότε θα ξανάρθω για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, το αντικείμενο, την ιδέα, το χρονοδιάγραμμα. Όλα μαζί θα τα συζητήσουμε και θα τα αποφασίσουμε. Ε, και θυμάμαι μερικές φορές από εκνευρισμό, ε, ε, μάλλον ε, ε, θυμάμαι που θυμώναμε όταν δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στους επιτρόπους αυτή, ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι βέβαια δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Να είναι σημαντικό να έχουμε επιτρόπους που να εκπορεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να συνεχίσω λίγο από εκεί, πολύ συγκεκριμένα. Σήμερα έχει οξυνθεί η κατάσταση με το Brexit θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών και να προσανατολισόμαστε εκεί. Και σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης, ποιο μηχανισμό θα χρησιμοποιήσετε μετά το Brexit για τους πολίτες στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι 1,8 εκατομμύρια και ε, έχουν αξίωση και δικαιούνται να έχουν Ιρλανδική υπηκότητα, άρα να είναι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να τους εξασφαλίσετε ένα δρόμο επιστροφής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείω διαφορετική ερώτηση, αλλά ναι, ας μιλήσουμε για την ε, ηθαγένεια. Ε, όπως ε, ξέρετε, όλες οι συμφωνίες απόσυρσης και αυτά που είχαμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο στην περασμένη θητεία, ανέκαθεν ναι, βάζαμε την ηθαγένεια στο πρώτο σημείο στην μερίσια μας διάταξη. Είδατε στην τελευταία σύσταση για αυτή την Επιτροπή έστειλαν επιστολή στα 27 κράτη-μέλη και είπαν ας είστε γενναιόδοροι αν δεν υπάρξει συμφωνία. Εγώ ελπίζω πως θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Η Ιθαγένεια λοιπόν είναι πολύ σημαντική, ειδικά όταν μιλάμε για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία και πρέπει αυτό το ζήτημα να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Γενεοδορία βέβαια δεν θα αρκέσει, θα πρέπει να κάνουμε κάτι, περισσότερο. Τόσο για τους Βρετανούς πολίτες εδώ στην Ευρώπη, όσο και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ε, στα Βρετανικά νησιά. Thank Σας ευχαριστώ, γιατί για το Ευρωκοινοβούλιο αυτό το σημείο για τη δική μας Επιτροπή τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών πολιτών που ζουν στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό σημείο. Τώρα ξεκινάμε το δεύτερο γύρο. Έχουμε 18 ε, ομιλητές ε, που προέρχονται από την Επιτροπή Γυναικών Απασχόλησης επίσης. Πρώτος ο κύριος Βίτσικ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σα, υποψήφια Αντιπρόεδρε. Σα ευχαριστώ για τι απαντήσει σα μέχρι τώρα και για την εισηγήσή σα, καθώ και για τι γραπτέ σα απαντήσει. Παρόμοιες ερωτήσεις ε, όλοι κάνουμε. Ε, ε, τι θα είναι αυτή η συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, ρωτάμε. Με άλλα λόγια ο καθένας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Μιλήσατε για το ρόλο του και τις σχέσεις με την Κομισιόν και το Εποπτικό Συμβούλιο, αλλά πιστεύω πως πραγματικά πρέπει να φτάσουμε στα κράτη-μέλη. Και με χαρά άκουσα τη δέσμευσή σας ότι επισκοπεύετε να επισκεφτείτε όλα τα κράτη-μέλη διερωτώ αν θα ε, απαιτήσουμε, απαιτήσετε την ίδια δέσμευση και από τους υπόλοιπους επίτροπους. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να μπούμε και να ε, επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή στις τελευταίες ευρωεκλογές αλλά είχαμε και κάποιες ε, αποτυχίες όπως στη δική μου χώρα που πολύ λίγοι ε, πολίτες πήγαν να ψηφίσουν. Ευχαριστώ. Ξέχασα να πω ότι πρόκειται για μία από τις ε, βασικές πολιτικές προτεραιότητες και κατευθυντήριες γραμμές της υποψήφιας Προέδρου. Πρέπει να επισκεπτόμαστε, να επισκεφτούμε μάλλον όλα τα κράτη-μέλη στο πρώτο τμήμα της θητείας. Και αυτό ισχύει για όλους τους επιτρόπους και για μένα ίσως περισσότερο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα επισκεφθούμε τα κρατημέλη, θα συζητήσουμε μαζί τους, θα τα ακούσουμε. Να επισκεφτούμε τα κρατημέλη δεν σημαίνει να επισκεφτούμε μόνο το κοινοβούλιο. Φυσικά θα το επισκεφτούμε και θα έχουμε συζητήσεις με τους βουλευτές, αλλά επίσης και έξω από τις πρωτεύουσες θα πρέπει να βρεθούμε, γιατί ο διάλογος με τους πολίτες γίνεται, αλλά συνήθως στις πόλεις και στις ε, μετροπολιτικές περιοχές, στα αστικά κέντρα. Θα πρέπει να βγούμε από αυτές τις περιοχές, να συζητήσουμε και με τους πολίτες εκτός, στην Ήπεθρο. Θα είναι ίσως διαφορετικό. Δεν λέω πως η τωρινή Επιτροπή δεν το έκανε, αλλά πρέπει να το τονίσουμε, να διευρύνουμε αυτή την δραστηριότητα, να δούμε ποιες είναι οι ανησυχίες των πολιτών μας. Αυτή θα είναι η δουλειά μου, αν φυσικά με επιβεβαιώσετε, με γκρίνετε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ακούω πως δεν θα βασιστούν όλα μόνο στις Βρυξέλλες, γιατί πιστεύω πως θα πρέπει να φτάσουμε τους πολίτες, αλλά και έξω από τα σύνορα της Ένωσης. Στην ομιλία σας λέτε ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους, ε, τον υπόλοιπο κόσμο για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ε, λειτουργεί και ποια είναι τα αποτελέσματα. Πώς λοιπόν θα παρουσιάσετε την Ευρώπη και στις υποψήφιες χώρες, ώστε και εκείνες να έχουν ε, τη, ε, λόγο για το μέλλον τους. Ίσως ε, σε επόμενα, στα επόμενα λίγα χρόνια μπορεί να μειωθούμε τα κρατημέλη, αλλά μπορεί και να πολλαπλασιαστούμε. Στο παρελθόν, ε, στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης υπήρχε χώρος για τα ε, χώρες της ε, διεύρυνσης. Πώς λοιπόν θα έχουν λόγο και τα κράτη-μέλη με τα οποία γίνονται ενταξιακές διαπραγματεύσει, γιατί και εκείνοι θα πρέπει να έχουν λόγο για το μέλλον του. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σα, κύριε Βλάτστικ. Ε, θα πρέπει να γνωρίζετε πω είμαι υπέρ τη διεύρυνση. Προέρχομαι εξάλλου από μια χώρα που ε, ενδιαφέρθηκε πολύ για τη διεύρυνση. Όμω, για αυτήν την ε, φορά θα γίνουν διάφορες συνελεύσεις σε διαφορετικά πλαίσια. Δεν θα συμπεριληφθούν στην, στην πρώτη συνέλευση. Πρώτα πρέπει να καθορίσουμε το δικό μας μέλλον, αν και μπορεί να φανεί κάπως αλαζονικό ε, προερχόμενο από μένα που είμαι από μια χώρα που ε, εντάχθηκε από τις τελευταίες στην Ένωση. Αλλά πάντως σε αυτή τη συνέλευση δεν θα συμπεριληφθούν τα ενταξιακά τα, τα κράτη αυτά γιατί εδώ θα μιλήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Ξέρετε ότι το μέλλον της Ευρώπης συζητήθηκε και από τους πρωθυπουργούς στο Στρασβούργο και μόνο από εκείνους. Αλλά σίγουρα οι συνομιλίες με τις υποψήφιες χώρες θα γίνουν αλλά με διαφορετική μορφή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρμπετ τώρα μάλλον στον σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ. Κυρία υποψήφια πρόεδρε, είναι σημαντικό να έχουμε ε, μια διάσκεψη με ευρυφάσμα συμμετεχόντων. Έτσι όμως αναφυσβήτα θα ε, ε, συναντήσετε κάποιους πολιτικούς που εσκεμένα κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσει, παραπληροφορούν ε, και ψεύδονται ή εξαπατούν τον κόσμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Αντίστοιχη πρόκληση αντιμετωπίζαμε στο Βρετανικό δημοψήφισμα και συνεχίζει αυτή η κατάσταση και στις ε, σημερινές συζητήσεις. Εσείς, στα πλαίσια της εντολής σας, τι πρόκειται να κάνετε για να βελτιώσετε την ενημέρωση και την γνώση της κοινή γνώμης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη αυτή τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη, αλλά και καλύτερη ενημέρωση του κοινού για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ. Σα ευχαριστώ κύριε Κόρμπετ. Όντω, είναι δύσκολο να εμποδίσουμε κάποιον, να τον αποτρέψουμε από το να μιλάει. Είμαστε ανοιχτή κοινωνία, ανοιχτέ κοινωνίε και ο καθένα έχει το δικαίωμα και την ελευθερία έκφραση. Φυσικά δεν είμαστε υπέρ τη παραπληροφόρηση ή ε, της διάδοσης ψευδών ειδήσεων ή παραπλανητικών πληροφοριών, αλλά είναι δύσκολο να το αποτρέψουμε, γιατί υπάρχουν πολλοί και διάφοροι πολιτικοί και μερικοί προσπαθούν ε, απλώς να, για ψηφοθυρικούς λόγους να ε, πείσουν τους πολίτες και δεν μπορούμε να τους βουλώσουμε το στόμα. Πάντως υπάρχει πρόβλημα. Στην παρούσα κατάσταση έχουμε κάποιους πολιτικούς που όταν γυρίζουν στην πατρίδα τους κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι είναι υπέτεια για το α το β, ενώ όταν ε, έρχονται στις Βρυξέλλες όλα τα βρίσκουν ωραία. Οπότε ε, έχουν αυτή τη προσωπία. διαφορετική συμπεριφορά ε, όταν είναι στην πατρίδα τους και διαφορετική όταν είναι στην Ευρώπη. Και αυτοί είναι που διασπείρουν αρνητικές ειδήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, έντιμοι και ειλικρινείς και να μιλούμε στον κόσμο. Αλλά δεν βλέπουμε τι μέσα θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τη σωστή ενημέρωση. Γιατί όντως κάποιοι δικοί σας συμπατριώτες προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο και αρχίζουν και το καταφέρουν με το λαϊκισμό, με τη δημαγωγία. Αλλά δεν θέλω τώρα να εμπλακώ ή να παρέμβω σε εσωτερική πολιτική συζήτηση. Οπότε βάζω τελεία εδώ. Γιατί, γιατί να σταματήσετε. Εσείς αν είχατε τον Πρωθυπουργό μιας χώρας μέλος που ήταν η βασική πηγή παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων, εσείς πώς θα το αντιμετωπίζατε, αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργό μιας χώρας ήταν ο αυτούργό τέτοιων παραπληρο, παραπλανητικών πληροφοριών. Ναι, όντω. Ε, Μερικέ φορέ το κάνουν ακόμη και πρωθυπουργοί, αλλά είναι ελεύθεροι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Μέχρι ότου του πιστέψουν οι πολίτε. Εκτό μικροφώνου, δυστυχώ, στα σχόλια του κ. Κόρμπετ. Διαφωνώ, δεν είναι καλό το ψέμα, αλλά είναι δύσκολο να το σταματήσουμε. Γιατί σήμερα έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα είναι ανοιχτά, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ο πολίτης θα κρίνει αν θα πιστέψει αυτό που ακούει ή όχι. Θα είναι δύσκολο να το σταματήσουμε αυτούς τους πολιτικούς. Πάντως, με τη διάσκεψη της Ευρώπης θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Και γι' αυτό θέλουμε να πλησιάσουμε τους πολίτες. Και γι' αυτό η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα γίνει. Είναι ένας από τους λόγους. Να έρθουμε κοντά στους πολίτες, να τους πλησιάσουμε. Και ήταν ιδέα βέβαια αρχικά του Πρόεδρου Μακρό, αλλά τη δεχτήκαμε όλοι. Την αισθανιστήκαμε όλοι, γιατί είναι καλό να μιλήσουμε με τους πολίτες. Πολλοί μιλούν για τη φούσκα των Βρυξελών, για το μικρό κόσμο αυτό που είναι απο, απομονωμένος, αποκομμένος. Εμείς θέλουμε όμως να φτάσουμε στον κόσμο και να συζητήσουμε με τους πολίτες, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του διαδικτύου. Η κυρία Ζαχαροπούλου από το Renew Europe, που είναι μέλος της Επιτροπής των Γυναικών, θα θέσει την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Όταν κανείς προβληματίζεται για τη δημογραφική μετάβαση, ασχολείται βέβαια και με τη γύρανση αλλά και με τη γεννητικότητα. Ε, σήμερα σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν πολιτικές γεννήσεων που προβλέπουν ε, επιδόματα γεννήσεων ε, εφόσον παραμένει παραδοσιακή εικόνα της οικογένειας. Αυτό παραγνωρίζει την έννοια της σύγχρονης οικογένειας με την πολυμορφία της, αλλά επιπλέον εισάγει διακρίσεις, στιγματίζει τις γυναίκες που θέλουν ή δεν θέλουν να έχουν παιδιά. Η δημογραφία δεν μπορεί να στρεβλώνεται ούτε να χειραγωγείται εις βάρος των ε, γυναικών. Ελπίζω αυτό να μην το υπονοεί ο τίτλος του ε, χαρτοφυλλοκίου σας. Ε, τι γνώμη έχετε για αυτές τις αρχαϊκές πολιτικές γεννήσεων και πώς θα αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική μετάβαση με τις σημερινές οικογένειες, τις οικογένειες του σήμερα που είναι πάρα πολύ ποικίλε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Σίγουρα είμαι πεπισμένη ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό δεν πρόκειται να τύχει κατάχρηση προς την κατεύθυνση που αναφέρετε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ε, δεν συζητούμε καθόλου το δίκτυο των γεννήσεων, σε καμία περίπτωση. Η οικογενειακή πολιτική μπορεί να είναι σημαντική, αλλά εξαρτάται από τον ορισμό της οικογένειας. Ε, δεν ε, θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά ε, η εξισορρόπηση του επαγγελματικού με τον ε, οικογενειακό βίο είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό είναι τμήμα του χαρτοφυλακίου μου και του χαρτοφυλακίου μου. Αν ακούσατε προσεκτικά, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο έχουμε την προστασία των παιδιών, έχουμε την ισορροπία του επαγγελματικού με τον ιδιωτικό βίο και τη γύρανση. Συμπεριλαμβάνονται λοιπόν οι πάντες και η ύπεθρος. Καμία σχέση λοιπόν με αυτή την συντηρητική ε, προσέγγιση και τους συντηρητικούς ορισμούς της δημογραφίας. Και θα μπορούσα ίσως να προσθέσω ακόμα το εξής. Ό,τι και να κάνω θα γίνει μετά από χαρτογράφηση. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία της Eurostat και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε. Ό,τι κάνουμε θα είναι με βάση στοιχείων και δεδομένων. Και δεν πρόκειται να προωθήσουμε καμία νομοθεσία χωρίς να έχουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που θα μας δίνει η Eurostat. Η κυρία Ζαχαροπούλου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Με ικανοποιεί ε, που σας ακούω να μιλάτε για ένα νέο ορισμό της οικογένειας, γιατί ως Ευρωβουλευτής ήσασταν αντίθετοι με τα δικαιώματα των γυναικών, ιδιαίτερα με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική ε, υγεία και κατά των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Και ως Επίτροπος Δημογραφίας θα πρέπει να συνεργάζεστε με την Επίτροπο ε, για ε, την Υγεία και την Επίτροπο για την Ισότητα που τάχτηκαν και οι δύο υπέρ των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ. Εάν συνεργαστείτε, πώς θα συνεργαστείτε με τις δύο συναδέλφους σας για να έχετε όλες ένα κοινό όραμα να προωθείτε. Thank you for your next... Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, προφανώς. Θα συνεργάζομαι και θα επικοινωνώ με όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα με τη συνάδελφο που είναι αρμόδια για θέματα ισότητας, την κυρία Ντάλη, Οπωσδήποτε θα είμαστε σε επικοινωνία, αλλά όπως σας είπα, ε, ε, είναι συλλογικό σώμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διέπεται από συλλογικότητα. Ε, ό,τι κάνουμε βεβαίως θα είναι προοδευτικό και θα είμαστε αρκετά προοδευτικοί για να προστατεύουμε τους πάντες. Η μη διακρίση είναι ένα στοιχείο ε, που είναι κατοχυρωμένο στι συνθήκε. μην αμφιβάλλετε. Αναφερθήκατε σε μου στάσει σε ψηφοφορίε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα ποτέ με το φύλλο ή τα δικαιώματα των Ε Πάντα ήταν δημοσιονομικοί οι λόγοι ή κάτι τέτοιο οικονομικό που μας έκαναν εκείνη τη στιγμή να μην μπορούμε να δεχθούμε ε, κάποια θέματα. Δεν έχουν να κάνει τα δικαιώματα του φίλου. Πάντα είμαι υπέρ ως γυναίκα, έχω και μια κόρη, έχω δύο εγγονές. Πώς είναι δυνατόν να είμαι κατά των δικαιωμάτων αυτών που συνδέονται με το φίλο; Μιλήσατε για τους ΛΟΑΤΚΙ. Και αυτό είναι η διάκριση. Σήμερα ε, εάν κάποιο στρέφεται κατά των δικαιωμάτων του, βεβαίω αυτό είναι στάδια Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τι προσωπικέ μου πεπιθήσει. Ε, πάντα θα πριτανεύει η συλλογικότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. E Τώρα ο κύριο Στεχόφσκι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε, το 2017 το 19% του πληθυσμού μας ήταν άνω των 65 ετών. Ερώτησή μου είναι, επειδή το χαρτοφυλάκιό σας ε, περιλαμβάνει την γύρενση και τους ε, ηλικιωμένους πολίτες, η ερώτησή μου είναι λοιπόν πώς σκοπεύετε να ε, εμπλέξετε αυτή την ομάδα ανθρώπων σε πιο ενεργή ζωή. Πολλοί πιστεύουν σε αυτές τις ηλικίε ότι υπάρχουν πολλοί φραγμοί που τους εμποδίζουν από την πλήρη τους ε, ανάμειξη στην καθημερινή ζωή. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω διπραγματεύσει με τα κράτη-μέλη, γιατί ίσω αυτό να μην είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ασχοληθούμε περισσότερο όμω με αυτό το θέμα για να βελτιωθεί η θέση των ηλικιωμένων στην κοινωνία μα. Ευχαριστώ, Τόμας, για αυτή την ερώτηση. Όπως είπα στην αρχή, ζούμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία. Είναι υπέροχη ευκαιρία και πρέπει να το γιορτάσουμε αυτό, αλλά είναι και πρόκληση για την κοινωνία, όπως ξέρετε. Μπορεί αυτό να είναι πρόβλημα για την συντάξη, για τα συστήματα συντάξεων, για το σύστημα υγείας ε, και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε ε, τους ηλικιωμένους στην κοινωνία. Υπάρχει μια ε, σημαίνια οικονομία που θα μπορούσε να... Ε, ανθίσει. Υπάρχουν πολλά, πολλοί τρόποι που μπορούμε να αναπτύξουμε μαζί, ώστε οι ηλικιωμένοι να αισθάνονται δραστήριοι. Και αυτή είναι η ιδέα με την οποία ασχολείται και η Γενική Διεύθυνση Επασχόλησης και η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Thank you very much for concrete answer. Ευχαριστώ για τη συγκεκριμένη σας αυτή απάντηση. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την ε, μέρημνα για τα παιδιά και τα δικαιώματα των παιδιών. Η ερώτησή μου είναι πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ευρώπη, όπου ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες, όπου τα παιδιά ε, ε, μπορεί να τα πάρουν από, τα από τους γονείς τους και να τα δώσουν σε στετούς γονείς. Μιλώ για το σκάνδαλο της Νορβηγίας και τον Μπάρτε Μπέρεντ, όπου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ε, ε, γίνονται πολλά εντελώς απαράδεκτα πράγματα και όπου πρέπει να τα συζητήσουμε με τους Νορβηγούς φίλους και εταίρους. Ε, ευχαριστώ. Τόμας, δεν τη γνωρίζω αυτή την υπόθεση, αλλά ό, όταν μιλάς για το χαρτοφυλάκιό μου και την προστασία των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου μου. Ε, η γύρανση, τα παιδιά, τα δικαιώματα των παιδιών, η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής και μάλιστα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας για την εγγύηση για τα παιδιά. Εργάζομαι για αυτήν την εγγύηση για τα παιδιά μαζί με τον Επίτροπο Σμιτ. Πολύ σημαντικό μέσο που θα μεριμνήσει για τα παιδιά. Είναι σήμερα ε, το 1 τέταρτο των, Ευρωπαίων, των παιδιών της Ευρώπης ζουν ε, στη φτώχεια. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αναπτύξουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Μια Πέτρα Κουπουλανάτρη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Σουίτσα, υποψήφια από την πανέμορφη Κροατία. Πολύ καλές ιδέες ακούσαμε για την διάσκεψη ε, και τη συνεργασία σας με, το, με την Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα η δημοκρατία δεν είναι μόνο πάμε και ψηφίζουμε, αλλά μια κοινωνία συμμετοχική, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε ο καθένας να μπορεί να διαβιώνει και να συμμετέχει στη δημοκρατία, άσχετα από πού προέρχεται, από την πεποίθησή του, από ποιον, ποιον ερωτευμένος, με ποιον ζει και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί πολίτες νιώθουν ότι τους μπρώχνουμε στο περιθώριο και αυτό τροφοδοτεί κάποιες ε, λαϊκιστικές ε, τάσεις και συγκρουσιακό κλίμα εις βάρος των μειονοτήτων και των γυναικών. Μερικές φορές φοβούμαι ότι πολυδρομούμε στην Ευρώπη. Ένα από τα βασικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου σας είναι να μεριμνήσετε ότι όσοι νιώθουν ότι έχουν μείνει πίσω να βοηθηθούν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Ε, και το άρθρο 2 του βιβλίου που μας δείξατε αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των, δικαιω... των δικαιωμάτων ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Πώς λοιπόν θα συμπεριλάβουμε καλύτερα, θα ενσωματώσουμε καλύτερα τις μειονότητες στην κοινωνία και τη δημοκρατία μας. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ σημαντική. Και το, κορτο, το χαρτοφυλάκιό μου και οι πολιτικές κατευθύνσεις της Νέας Επιτροπής μιλούν για συμμετοχή, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό είναι το κλειδί για μας. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε τους πάντες. Και όταν μίλησα για μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για Ευρωπαίους πολίτες, είχα στο μυαλό μου και τις μειονότητες. Φυσικά και οι μειονότητες είναι σημαντικές. Είναι σημαντικό της κοινωνίας μας και πιστεύω στην, και στη δική του συμμετοχή. Σε καμία περίπτωση δεν θα περιθωριοποιηθούν οι μειονότητε, δεν θα αποκλείσουμε κανέναν. Και είπατε για αυτού που υστερούν, που έχουν μείνει πίσω. Ε, όταν μιλούμε όμω για ανθρώπου που έχουν μείνει πίσω, ε, είναι κυρίω αυτοί που μένουν είτε στην ύπεθρο στι αγροτικέ περιοχέ, είτε σε κάποιε ε, περιφέρειες τη Ευρώπη ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε ε, μεγάλες ε, μεταναστευτικές ροές, δημία τοπικού πληθυσμού, διαρροή εγκεφάλων, ε, γιατί οι καλύτεροι φεύγουν. Οπότε ο κόσμος νιώθει αποξενωμένος, νιώθει ότι τους έχουν αφήσει πίσω και δεν θέλουν πια να συμμετέχουν, γιατί η δημοκρατία σημαίνει και συμμετοχή. Γι' αυτό και έχει σημασία να είμαστε ανοιχτοί προς τους πάντες για συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς. Πάντως να είστε ήσυχοι θα μεριμνήσουμε και για τις μειονότητες. Ε, λόγω εθνικής προέλευσης, πεπιθήσεων και ούτω Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλύψει τους πάντες. Άλλωστε δεσμευόμαστε και από τη συνθήκη το άρθρο 2 που επισημάνατε. Αλλά δεν το λέω μόνο επειδή το γράφει η συνθήκη, είναι και προσωπική μου πεποίθηση η συμμετοχή χωρί αποκλεισμού. Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία για τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη ε, στηρίζεται στην αρχή ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να συμμετέχουν, να έχουν και αυτοί λόγο στην όλη διαδικασία. Υπόσχεστε ότι θα καλέσετε μη κυβερνητικέ οργανώσει, κοινωνία των πολιτών, νεολαία ή οργανώσει νεολαία, αλλά δεν θα αποκλείσετε ε, όσους εκπροσωπούν σεξουαλικές μειονότητες ή εκπροσώπους άλλων μειονοτήτων ή, μειονο... ή εκπροσώπους των οργανώσεων που ε, προστατεύουν ε, σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Γιατί θυμάμαι και την πρωτοβουλία για το δικαίωμα στην άμβλωση. Ε, δεν θυμάμαι να είστε και πολύ θετικοί. Εσείς ως Επίτροπος, αν εκλεγείτε τελικά, ποια θα είναι η στάση σας για τα θέματα αυτά. Καταρχήν, να αναφερθώ στην ψήφο μου και στην έκθεση πρωτοβούλες. Αν θυμάστε καλά, ήταν ε, μια έκθεση εφαρμογής μετά από ένα χρόνο εφαρμογής. Και ήταν πρόβλημα πάλι δημοσιονομικών πόρων, γι' αυτό και καταψήφισα τότε. Είχα υποβάλει εναλλακτικό ψήφισμα, αλλά αυτό δεν είχε καμία σχέση με τη θέση μου για τις μειονότητες ή για οποιοδήποτε ομάδα της κοινωνίας. Αλλά μου ζητήσατε να κάνω μία υπόσχεση. Στην προετοιμασία που μου έκανα μου είπαν μην δίνετε και πολλές υποσχέσεις. Ε, αλλά αυτό μπορώ να σας το υποσχεθώ, γιατί ούτως ή άλλως συνάδει με τις προσωπικές μου πεπιθήσεις. Μείνετε ήσυχοι. ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Φρόιντα από την ομάδα των Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Όταν σκέφτομαι το μέλλον της Ευρώπης, σκέφτομαι το Ζαν Μονέ, τον Αλτιέρο Σπινέλη, την Ούρσουλα Χίρσμαν, τη Λουίς Βάις και τις δικές τους αντιλήψεις για το μέλλον της Ευρώπης. Σκέφτομαι μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, γνήσιες ευρωπαϊκές εκλογές με υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Σκέφτομαι το κράτος δικαίου που θα προστατεύει τους πολίτες και όλες τις δυνατότητε τα ίσα δικαιώματα για άνδρες, γυναίκες, ε, για ε, ομοφιλόφιλους, ετεροφιλόφιλους. Σκέφτομαι θεσμικά όργανα διαφανή και αδιάφθορα η κυρία Φόντερ Λάιεν ε, υποτίθεται ότι θέλει να χτίσει την Ευρώπη στις ίδιες αρχές και αξίες. Εσείς όμως επανειλημμένα τα περασμένα χρόνια ε, καταψηφίσατε τη διαδικασία άρθρου 7 για την Ουγγαρία, καταψηφίσατε τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια, καταψηφίσατε την περισσότερη διαφάνεια στο Συμβούλιο και ε, τους ισχυρότερους κανόνες για τα λόμπι, για να σας αναφέρω ενδεικτικά και μόνο μερικά παραδείγματα τώρα σας έχει ανατεθεί μια αποστολή από την εκλεγμένη πρόεδρο. Πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτή και πώς είναι δυνατόν ε, αξιόπιστα να υπερασπίζετε το μέλλον της Ευρώπης που βασίζεται σε αυτές τις αξίες. Σήμερα θα ψηφίζετε διαφορετικά σε κάποια από αυτά τα θέματα. Απάντηση. Κύριε Φρόντ, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Εγώ πιστεύω στο κράτος δικαίου, πρώτα απ' όλα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, για να το εξηγήσω, που είναι το άρθρο 7. Είναι το πιο εύκολο αυτό να το εξηγήσω. Φυσικά και πιστεύω στο κράτος δικαίου. Αυτή η έκθεση σε Αρχεντίνη ήταν έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου και δεν μιλούσαμε για την Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι ένας ουδέτερος διαιτητής Γι' αυτό η δική μου αντιπροσωπεία καταψήφισε. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω. Φυσικά ανησυχώ όταν υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις του κράτους δικαίου εκεί και συμμερίζομαι την άποψή σας, αλλά εξ όσων γνωρίζω το θέμα εκρεμεί τώρα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, αλλά έχει... Ε, οδηγηθεί σε εμπλοκή στο Συμβούλιο. Βεβαίως και πιστεύω στο κράτος δικαίου, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφορές όταν ζεις σε μια χώρα όπως είναι η πατρίδα μου, η οποία συνορεύει με τη χώρα που αναφέρατε. Έχω πει και στο παρελθόν. Είναι πιο εύκολο να μην είσαι ευρωβουλευτής και να έρχεσαι στην ακρόαση του Επιτρόπου. Όπως σας είπα, η Ευρώπη διέπεται από συλλογικότητα. Αυτό το πνεύμα πριτανεύει. Ομόφωνα αποφασίζουμε και παρακαλώ να μην αμφισβητείτε ε, τις πεπιθήσεις μου και τις στάσεις μου σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια. Ε, Θα ήθελα να ε, συνεχίσω για το ρόλο που θέλετε να παίξετε στη διάσκεψη για την Ευρώπη. Την τελευταία θητή είχαμε πολλές εκθέσει στο Κοινοβούλιο, την έκθεση των πέντε προέδρων. Εσείς ίδια μιλήσατε για τους πολυπληθείς διαλόγους με τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διεξαγάγει. Περίπου 200.000 πολίτε συμμετείχαν άμεσα. Ε, όλοι οι ηγέτες, όπως είπατε, οι πρωθυπουργοί ήρθαν και εξέθεσαν εδώ την άποψή του στο Κοινοβούλιο και το όραμά Είναι τεράστιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη από την κλιματική αλλαγή ε, μέχρι τους μεγάλους ε, πολυεθνικούς ομίλους που δεν πληρώνουν φόρους στην Ευρώπη. Τι θα κάνουμε με την ψηφιοποίηση, ε, πώς θα υπερασπιστούμε το ρόλο της Ευρώπης σε έναν κόσμο ανάμεσα σε Ηνωμένε Πολιτείες και Κίνα. Έχει έρθει τώρα η ώρα να πάμε δύο χρόνια για να ακούμε, όπως λέτε τους πολίτες. Δεν έχει έρθει η ώρα για δράση και αν έχει έρθει η ώρα για δράση, ε, λέτε θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που δίνουν οι συνθήκες χωρίς να πάτε αμέσως σε τροποποίηση των συνθήκων. Μπορείτε να μας δώσετε τα τρία σημαντικότερα που θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία και μπορούμε να τα κάνουμε με τις κείμενες συνθήκες. Και ρωτώ τη δική σας προσωπική άποψη θέλω να έχω, όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που πιστεύετε εσείς έχει τώρα τη μεγαλύτερη σημασία. Μα, αφού με ρωτάτε τόσο ε, ε, ευθέω, θα απαντήσω ευθέω. Η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντικό θέμα και το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Τίμερμαν αυτή τη στιγμή είναι από τα σημαντικότερα. Αυτό ε, βλέπω έτσι, για το μέλλον της Ευρώπης. Αλλά φυσικά και η ψηφιακή μετάβαση είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να αρχίσουμε από αυτά. Αλλά γιατί να θεωρήσουμε τις συνθήκες για να δράσουμε. Μπορούμε να δράσουμε αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες που έχουμε. Είμαι υπέρ αν χρειαστεί, αν το δείξουν αυτό οι συζητήσει. Δεν θέλω να επιβάλλω τίποτα. Και είμαι βεβαία ότι ούτε η ε, εκλεγμένη αντιπρόεδρος θέλει να επιβάλλει κάτι. Για την τροποποίηση των συνθηκών θα την κάνουμε αν τη ζητήσουν οι πολίτες. Φυσικά εσείς είστε οι άμεσα εκλεγμένοι. Εμεί είμαστε οι άμεσα εκλεγμένοι ε, εκπρόσωποι των πολιτών. Φυσικά, το κλίμα και ε, η ψηφιακή Ευρώπη είναι τα σημαντικότερα και πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά με την αρχιτεκτονική που έχουμε και με τη συνθήκη που έχουμε. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση από την κυρία Φράνζα Με. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, απόψε μιλάμε για δημοκρατία και για δημογραφία. Τι να πούμε λοιπόν για τη λειτουργία αυτού του θεσμού που δεν επιτρέπει στους ε, λαούς, στους κυρίαρχους λαούς να αποφασίζουν για το δικό τους μέλλον μέσω ενός συστήματος που συγκεντρώνει τη δημοκρατία στις Βρυξέλλες. Και μιλώ για την Ουγγαρία και την Πολωνία που εκείνοι ε, θέλησαν να αρνηθούν την μετανάστευση που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και που σήμερα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ερώτησή μου λοιπόν, κυρία υποψήφια Επίτροπε, είναι κατά τη γνώμη μου η δημοκρατία δεν έχει νόημα παρά στο μέγεθος ενός κράτους ε, και ενός λαού. Θα αφήσετε λοιπόν τους λαούς να, να έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Και έπειτα, γιατί να μην ξεκινήσουμε μια πραγματική πολιτική υπέρ των γεννήσεων που να βασίζεται στην οικογένεια παρά να στηρίζουμε μια πολιτική υπέρ της μετανάστευσης. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Ζαμέ. Είπα στην αρχή ότι υπάρχει πάντοτε αντιπαράθεση ανάμεσα στην αντιπροσωπευτική και στην άμεση δημοκρατία. Θέλετε οι λαοί να αποφασίζουν. Οι λαοί μας εξέλεξαν εδώ, εμάς, εσάς και έτσι έχουν το λόγο τους. Αλλά συνειδητοποιούμε ότι δεν αρκεί. Θέλουμε να ακούσουμε τους λαούς και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στην μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια ή τη μία φορά κάθε πέντε χρόνια, ανάλογα με όταν μιλάμε για εθνικές ή ε, αυτοδιοικητικές εκλογές. Και τώρα με, με ρωτήσατε για τη δημογραφία, τα ποσοστά γεννήσεων. Δεν βλέπω να υπάρχει εδώ πρόβλημα. Όταν όμως μιλάτε για μετανάστευση, ό,τι είναι νόμιμο είναι αποδεκτό. Νόμιμη μετανάστευση τη δεχόμαστε. Ξέρω πως αναφέρεστε σε κάποιες χώρες που δεν επέτρεψαν, δεν δέχτηκαν τους μετανάστες και να σας πω για τη δική μου χώρα. Η χώρα μου ε, περικλείεται από φράχτες. Όλες οι χώρες εκτός από μας δεν επιτρέπουν στους μετανάστες να έρθουν. Είτε είναι νόμιμοι είτε είναι παράνομοι. Καταλαβαίνω λοιπόν το τι λέτε, αλλά θα μπορέσουμε και αυτό να το συζητήσουμε στο πλαίσιο της συνέλευσης. Θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα θέμα για τη συνέλευση. Επερώτηση. Ναι, ε, μιλάμε εδώ και ώρα για τις, τα μεγάλα θέματα και θέλετε να βάλετε τους πολίτες στο επίκεντρο της συζήτησης. Να θυμίσω όμως ότι όταν οι Ιρλανδοί ψήφισαν όχι, τους ζητήθηκε να ξαναψηφίσουν. Όταν οι Ελβετοί ψήφισαν για τη μετανάστευση, τους ανάγκασαν μετά όταν ε, ε, η Ισλανδία αποφάσισε να μην μπει στην Ένωση, ε, ε, τους κυνηγάμε. Λοιπόν, άρα τι, πού είναι η δημοκρατία. Ε, ποια είναι η πραγματική δημοκρατία. Όταν ακούσουμε λοιπόν ε, τις απόψεις των λαών, πότε θα σεβαστούμε τις απόψεις αυτές, την ελευθερία τους και πότε θα σεβαστούμε εδώ ακριβώς την δημοκρατία. Θα κατανοήσετε ότι δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω με όλους σήμερα. Με σας δεν συμφωνώ, γιατί ε, σας εξέλεξαν εσάς και οι ψηφοφόροι σας αντέδρασαν μέσω του προσώπου σας και όχι μόνο οι ψηφοφόροι σας, αλλά μισό εκατομμύριο Μισό ε, ε, κάτοικοι είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες και εσείς εκπροσωπείτε τις απόψεις εκείνων που σας ψήφισαν και όλοι μας εκπροσωπούμε όσους μας ψήφισαν. Εκπροσωπούμε κάθε έναν Ευρωπαίο πολίτη που είναι άνω των 18 ετών ή των 16, ανάλογα με τον εκλογικό σας νόμο. Ε, ο Χέλμουντ Γκόκινγκ είναι ο επόμενο μιλητή από την ομάδα <laughs> ECR. με ευχαριστώ πολύ για όσα είπατε μέχρι τώρα. Δουλεύετε με τη Eurostat, λέτε, για τη δημογραφική αλλαγή. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι μεγάλη η πρόκληση. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την επικουρικότητα δεν θα πρέπει να έχουμε όλες τις απαραίτητες ε, στατιστικές για την οικογένεια, για τη φύλαξη των παιδιών, για τον ιδιωτικό και τον επαγγελματικό βίο. Τα περισσότερα δεδομένα θα έδειχναν ότι ε, στην Ευρώπη ε, εξαπατάμε τον κόσμο. Μεγαλώνουν παιδιά για να είναι φτωχοί γέροι μετά. Ποιες είναι οι λύσεις που θα προτείνετε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την δημογραφική αλλαγή, να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των ηλικιωμένων και να ενισχύσουμε κυρίως την οικογένεια. Αυτό θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Thank ευχαριστώ. Uh, Είπατε ό,τι ακριβώς θα κάνω στη δημογραφία ε, θα στηρίζεται στα στοιχεία της Eurostat. Θα εξαρτηθεί από το τι στοιχεία έχουμε. Όσα δεν έχουμε θα προσπαθήσουμε να τα συμπληρώσουμε. Θα κάνουμε μια χαρτογράφηση και θα δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Και με βάση αυτά τα στοιχεία και δεδομένα θα ξεκινήσουμε το έργο μας. Με βάση την επιστολή ανάθεση καθηκόντων, έχω το καθήκον μέσα στο πρώτο εξάμεινο να κάνω αυτή τη χαρτογράφηση τον απολογισμό της κατάστασης για να δούμε τι, πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Αυτή θα είναι η πρώτη έκθεση που θα εκπονήσω το πρώτο εξάμεινο. Με βάση τις επαφές μου με τη Eurostat γνωρίζω ότι έχουν πολύ αξιόπιστα και έγκυρα στοιχεία και μάλιστα έχουν αλλάξει και την προσέγγισή τους για την ε, συγκέντρωση αυτών των στοιχείων. Οπότε ο νέος κανονισμός πλαίσιο για τα κοινωνικά στατιστικά στοιχεία θα εμπλουτίσει τη βάση των πληροφοριών. Αυτά για τα δεδομένα και τη Eurostat. Σε ό,τι αφορά τώρα την καταπολέμηση της φτώχειας, όπως είπα και προηγουμένως, η γύρανση είναι πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Η συμφιλίωση ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου το ίδιο, πολύ σημαντικό. Και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα δούμε ποιε είναι οι δράσει των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολλέ αρμοδιότητες είναι εθνικέ. Εκεί που είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη, εμείς απλώς θα συνδράμουμε και θα δούμε μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τι μπορούμε να κάνουμε, είτε μέσω συστάσεων, είτε χρησιμοποιώντας άλλα μέσα. Ευχαριστώ. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Ζητώ συγγνώμη αλλά είναι πολύ λίγα αυτά που μας λέτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει το πλαίσιο και είναι και ευθύνη της. Και σας ερωτώ συγκεκριμένα. Ε, θα είστε υπέρ ενός ε, επιπλέον επιδόματος τέκνων και επιδόματος ανατροφής όπως υποστηρίζει το δικό μας κόμμα για τις οικογένειες στη Γερμανία. Θα δημιουργήσετε εκείνες τις προϋποθέσεις και το θεσμικό πλαίσιο για τους ανθρώπους όπως είπατε και ίδια προηγουμένως, το 25% των παιδιών, το 1 τέταρτο στην Ευρώπη ζουν στη φτώχεια. Πού είναι η ισότητα των ευκαιριών για την καινοτομία, για την εκπαίδευση. Χρειάζεστε γι' αυτό αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα. Για μας η Eurostat δεν επαρκεί. Ποιες άλλες αντικειμενικές πηγές ε, θέλετε να συμβουλευτείτε για να πάρετε στοιχεία και να τα συνυπολογίσετε. Για μας δεν αρκεί η Eurostat για να σας δώσει πληροφορίες. Πολύ συγκεκριμένα έχετε να μας πείτε άλλες πηγές αντικειμενικές τις οποίες θα προσφύγετε εκτός τη Eurostat. Αν θυμάστε, Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Πυλώνας είναι πολύ σημαντικός. Και όπως σας είπα, όταν υπάρχουν εθνικές αρμοδιότητες, τις σεβόμαστε. Θα πρέπει όμως να θεσπίσουμε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές και πρότυπα. Αυτό κάνουμε. Ο κοινωνικός πυλώνας προβλέπει 20 διαφορετικές δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν. Και περιλαμβάνει ε, αυτό και την συμφιλίωση ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου, την ε, διαβίου παροχή φροντίδας, τη διαβίου κατάρτιση. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα που έχουμε εγκρίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017. Ευχαριστώ. Η Κίνκα Γκάλ από το ΕΛΚ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Στην αρχική σας δήλωση, ε, που ήταν πολύ καλή, είπατε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δημογραφικές προκλήσεις. Ξέρω ότι στην Κροατία συμμετείχατε στην παρακολούθηση και εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την προστασία των οικογενειών. Θεωρείτε ότι η ανάπτυξη ε, ε, πολιτικών ε, υπέρ της οικογένειας θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Κίνγκα, για την ερώτησή σου. Γνωρίζουμε ότι συρρυκνώνεται το εργατικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπα και προηγουμένως αν παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση, εάν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις της μείωσης, το 2070 θα έχουμε χάσει 10% του εργατικού μας δυναμικού, αν παραμείνουν ε, οι γεννήσεις στα ίδια επίπεδα. Οπότε ο λόγος μεταξύ των όσων βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία και των συνταξιούχων θα επιδεινωθεί. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Οπότε αν έχουμε φιλοοικογενειακές πολιτικές σίγουρα θα παίξουν κάποιο ρόλο. Και μίλησα για τη συμφιλίωση ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου και φυσικά εννοείται ότι θέλουμε και φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές. Μόνο έτσι θα διευκολυνθεί ο συνδυασμός ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Θέλουμε καλύτερο άλλα εργασία, καλύτερες υποδομές για τους γονείς. Θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες ε, για να απασχολούνται περισσότερο, χάρη στους βρεφονιπιακούς σταθμούς που θα έχουν, χάρη στη φροντίδα των παιδιών που θα εξασφαλίζεται. Υποδομές που θα φροντίζουν την οικογένεια, φιλοοικογενειακές πολιτικές που θα διευκολύνουν το συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Αυτά είναι και βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα. Επερώτηση καλό θα ήταν να έχουμε τις ε, θετικές πρακτικές των κρατών μελών ε, για τις φιλοοικογενειακές πολιτικές και τις υποδομές φροντίδας των παιδιών, αν έχουν αποδείξει την αξία τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει κάποια κονδύλια. Μέχρι στιγμής 2,2 δισεκατομμύρια δαπανήθηκαν για τέτοιου είδους φιλοοικογενειακές πολιτικές, για τη διαβίου παροχή φροντίδας, και για αντίστοιχες πολιτικές. Και φυσικά είμαι υπέρ και της αγοράς εργασίας και υπέρ της εντονότερης παρουσίας των γυναικών στην αγορά εργασίας και την καλύτερη τους ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει καλές υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών τους. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μαϊτέ Παγκαθαουρτουντούα. Το Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Ταγιάννη. Η δημοκρατία. Η δημοκρατία αποτελείται από ε, το κράτος, δημοκρατικό κράτος δικαίου. Βασίζεται σε κανόνες, σε νόμους, ε, στην αρχή ότι ο πολιτικός πλουραλισμός είναι αυτοί οι πυλώνες που μας προστατεύουν από τα απολυταρχικά κράτη. κράτη. Ακριβώς για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιούργησε το άρθρο 2 και το 7, γιατί εφόσον υπάρχει ε, κίνδυνο σαφή να γίνει ε, ανελεύθερο ένα κράτος, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσουμε και να, για να προστατευτούμε. Και υπάρχει το άρθρο 7. Είναι ένα άρθρο υποστήριξη ε, του κράτου δικαίου. Ε, δυστυχώς στην Ουγγαρία ο κίνδυνο είναι η χώρα αυτή να γίνει ανελεύθερη και υπερεθνικιστική και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό. Thank you for your uh, This is very... Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας που είναι πολύ σημαντική και είμαι βεβαία ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει ε, δεν ότι τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη συνθήκη. Τα άρθρα αυτά θα πρέπει να τηρηθούν. κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μεριμνήσουμε και να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου όπως είπα σε μια από αυτές τις ε, χώρες υπήρξε σοβαρή ρήξη του κράτους δικαίου, παραβίαση μάλλον του κράτους δικαίου και συμμερίζομαι τις ίδιες ανησυχίες με σας, Αλλά νομίζω πως αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, όπως σας είπα είναι στο Συμβούλιο, να δούμε τι θα πει το Συμβούλιο, αλλά αυτό είναι ένας από τους λόγους όπου πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για ειδική πλειοψηφία. Έχετε επερώτηση. Ναι, βεβαίω. Η δεύτερη αφορά τη δημογραφία. Κοιτάξτε, εγώ έχω... Με απασχολεί πολύ η η κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ισπανία. Στο Βούργος ο δήμαρχος του Καλδαρών έχει 30 κατοίκους μόνο και μόνο και ένας από τους καλύτερους επιχειρηματίες κρασιού που γνωρίζω ζει στην Ήπεθρο και προσπαθεί να πουλήσει στο εξωτερικό το καταπληκτικό του κρασί. Ξέρετε τι λένε αυτοί οι φίλοι και άλλοι φίλοι που έχω στην τελείω αποψηλωμένη από ανθρώπους Ευρώπη, απεριμωμένη ότι χρειάζονται το ίντερνετ γιατί σε λίγο του χρόνου το Καλδαρόν θα έχει μηδέν κατοίκους. Θα μπορέσουμε να, να έχουν όλοι και στην Ήπεθρο ίντερνετ όπως έχουμε όλοι για να μπορέσει να αναπτυχθεί και η Ήπεθρος. Ναι, βεβαίως υπάρχουν περιφέρειες όπου δεν υπάρχει δίκτυο δεν υπάρχει ίντερνετ. Θυμάμαι σε μία από τις εκθέσεις της κατάστασης πρόοδου της Ένωσης είπε «Κάθε χωριό θα έχει Wi-Fi». Θα το θυμάστε νομίζω κι εσείς. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση, όπως ξέρετε, υπάρχει αυτή η έννοια το Wi-Fi για όλους ε, βελτιώνονται διαρκώς τα πράγματα, αλλά τώρα ξέρω πως υπάρχουν περιφέρειες που δεν έχουν ακόμα ίντερνετ, δεν έχουν ακόμα τις υποδομές. Γι' αυτό το λόγο όπως είπα, θα πρέπει να επισκεφτούμε όχι μόνο τις πρωτεύουσε, αλλά και τις περιοχές της υπέδρου. Πρέπει να φτιαχτούν οι υποδομές και γι' αυτό είπα ότι κλείνουν σχολεία, κλείνουν τα ε, ταχυδρομεία, ε, τα λεωφορεία δεν πάνε πια αλλά πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές. Μόλις θα φτιάξουμε τις υποδομές θα έχουμε το θέμα των θέσεων απασχόλησης. Υπάρχει μια πόλη στην Κροατία, το Μπούκοβαρ, που ξαναχτίστηκε μετά τον πόλεμο εντελώ. Φτιάχτηκαν τα σπίτια, ήρθε το Wi-Fi, ήρθαν όλα, αλλά δεν είχαμε δουλειές για αυτόν τον κόσμο. Πολύ περίπλοκη υπόθεση λοιπόν. Ο Επίτροπος για τη Συνοχή η επίτροπο για τη Συνοχή θα είναι πολύ πολύ σημαντική και θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σε συνεργασία με τους συναδέλφους. Κατανοώ το πρόβλημα γιατί ξέρω πολλές περιοχές όπως η αυτή που αναφέρατε εσείς στην Ισπανία. Υπάρχουν πολλές σε όλη την Ευρώπη. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε τη χαρτογράφηση ε, της κατάστασης μέσα στους πρώτους έξι μήνες. Πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε αμέσως. Μάρτιν Σόνεμπον, μη εγγεγραμμένο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίσατε ορίσατε τον Μπράφκα. Εσ. Ε, προτινόμενη Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόλες ε, τις προσπάθειες και τις εντατικές τα τελευταία 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να μειώσει το κατόφλι της, όφιας, της φτώχειας κάτω από 25%. Πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν στην φτώχεια ή απειλούνται από αυτή. Αυτά τα λέει Eurostat. Εσείς αντίθετα είστε ένα παράδειγμα που μπορεί να δώσει ε, στους Ευρωπαίους ελπίδα. Πριν από 20 χρόνια ε, ήσασταν ε, δασκάλα και είχατε ένα σαραβαλάκι ρενό και 60 τετραγωνικά σπίτι σε μια παλιά πολυκατοικία. Τώρα έχετε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, βίλα, δύο σπίτια, δύο διαμερίσματα, ένα εξοχικό, 12 ε, μέτρα σκάφος και τρία αυτοκίνητα. Θα μοιραστείτε την πατέντα σας και τη συνταγή σας με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εμάς, ο Πρόεδρος. Δεν είναι δουλειά μας να συζητάμε για το παρελθόν και για τα χρήματα. Έχει έρθει στην Επιτροπή για άλλο λόγο. Ε, στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Έχετε ερώτηση επί του θέματος. We need, we need to know. Everybody is free, but this is... Εντάξει, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ε, ό,τι θέλει, αλλά ε, ε, δεν είναι εκτός θέματος η ερώτηση. Μπορώ να απαντήσω. Δεν με πειράζει. Γιατί όχι. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα θέματα. Η τελευταία πρότασή σας ποια ήταν, γιατί δεν την άκουσα. Ρώτησα αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τη μυστική σας συνταγή. Αυτή την πατέντα που έχετε βρει. Thank Ευχαριστώ κύριε Ζόνεμπορν. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και θα απαντήσω στα αγγλικά μέχρι τώρα τα γερμανικά. Καταρχάς, δεν μιλάτε για πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι αυτά γεγονότα. Εμπνέεστε από κάποια άρθρα λανθασμένα. Ψευδή θα κάνω ό,τι μπορώ να πετύχει η πορεία μου σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Αν μιλάτε για μένα και για πριν από 20 χρόνια, δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι του παρόντος ούτε στο ύψο των περιστάσεων και του σεβασμού του Κοινοβουλίου. Αν πω μαζί σα σε τέτοια συζήτηση για το που έμενα πριν από 20 χρόνια, έμενα στο Ντουμπρόβλινγκ με τον άντρα μου, στο σπίτι τη οικογένεια μου που είναι εμποροπλίαρχος, ε, σε φορτηγά τότε, χίδιν φορτίου, σε πλοία με κοντέινερ και πρόσφατα σε κρουαζιερόπλια και έβγαζε αξιοπρεπή μισθό αν επιθυμείτε να το μάθετε, αν θέλετε να ξέρετε, το πόθεν έσχες μου ανέκαθεν ήταν διαφανές, ανοιχτό και σύμφωνα με τους κανόνες του θεσμού που εργαζόμουν. Είτε ήμουν ε, δήμαρχος στο Ντουμπρόβνικ ή μέλος του Κρατικού Κοινοβουλίου, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δήλωση οικονομικών μου συμφερόντων είναι γνωστή και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε είναι διαφανές, νόμιμο και σύμφωνα με τους κανόνες πάντα και σύμφωνα με τις θυσίες που έκανε η οικογένειά μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει να είσαι καπετάνιος και να θαλασσοπνίγεσαι σε τέτοια καράβια, σε όλα τα πελάγια και τους ωκεανούς. Καλά, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός εδώ. Όλα είναι σωστά, είναι σύνομα και θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου που απορρέουν από την επιστολή ανάθεσης εντολής και να βοηθήσω ε, τους Ευρωπαίους πολίτες, εκείνους που έχουν ανάγκη, που ζουν στη φτώχεια και είναι απόκληροι να ζήσουν ε, αξιοπρεπείς ζωές. Και ε, πιστεύω ότι αυτή η πενταετία θα είναι αρκετή για να τους βοηθήσουμε. Please. Ich habe Έχω συμπληρωματική ερώτηση. Ρενό 4, είχατε Ρενό 9. You know what? Ξέρετε κάτι. Πλοίο ήτανε. Σας ευχαριστώ. And now... Κύριε Γκλουξμαν από τους σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ε, το πλεονέκτημα ήταν ότι θετεύσατε και ως ε, βουλευτής, ευρωβουλευτής και όπως και ο συνάδελφος Φρόιντ ασχολήθηκα με το παρελθόν σας εδώ, για το ιστορικό σας. μας δι... Μα προβληματίζει η ψήφο σα. Η έκθεση Αρχεντίνη μιλούσε για άνοιξη τη διαδικασία στο άρθρο 7 για την Ουγγαρία και την καταψηφίσατε. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά γιατί θα αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο τη δημοκρατία. Και σήμερα μα μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να είναι ουδέτερο διαιτητής. Δηλαδή θα είστε ουδέτεροι ως προς τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορείτε να μας υποσχεθείτε γιατί θα πρέπει να προσδιορίσουμε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις για την ικανότητά σας να δράσετε υπέρ ενός αποτελεσματικού άρθρου 7. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα σήμερα, να μην παραβιαστούν οι αρχές μας και όταν προτείνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει συνέχεια και να ακολουθούν ε, δράσεις. Έχετε αλλάξει γνώμες προς το άρθρο 7 γιατί είχατε καταψηφίσει τότε την έκθεση Αρχεντίνη. μάλλον δεν καταλάβατε αυτό που είπα πριν. Είπα ότι πιστεύω στο κράτος δικαίου και είπα ότι πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να είναι ουδέτερος α, ε, διαιτητής. Και αν με εγκρίνετε ως αντιπρόεδρος θα ακολουθήσω ό,τι αποφασίσει το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μην φοβάστε καθόλου λοιπόν, μην αμφιβάλλετε ούτε για την ψήφο μου ούτε για τις πεπιθείς μου. Το άρθρο 7 είναι σημαντικό. Θα δούμε τι θα πει και το Συμβούλιο και τι θα πει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και όταν το θέμα φτάσει και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι θα ευθυγραμμιστώ απόλυτα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Μια και θέλω να συνεχίσω και προηγούμενες ερωτήσεις, θα συνεχίσω την, έκθεση, ε, την ερώτηση του κ. Τουράν από το Ρινιού για τη θεωρία της αντικατάστασης. Μπορείτε όντως να καταδικάσετε τους ε, πολιτικούς ηγέτες και κυρίως την Ουγγρική κυβέρνηση και τον ε, Πρωθυπουργό που μιλά για αντικατάσταση του ευρωπαϊκού πληθυσμού από πληθυσμό που θα προέρχεται από μετανάστευση. Και επίσης ε, επερώτηση σε κάποια άλλη ερώτηση για το δικαίωμα στην άβλωση. Ποια είναι η άποψή σας για το δικαίωμα στην άβλωση και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ευχαριστώ για τις συμπληρωματικές σας ερωτήσεις. Δεν πρόκειται να καταδικάσω κανέναν, γιατί δεν είμαι σε θέση να στείλετε έψω να καταδικάσω κανέναν. Πάντως, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα ακολουθήσω τις πολιτικές κατευθύνσεις και το πνεύμα συλλογικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να διαχωριστώ. Επίσης, μιλήσαμε για τη μετανάστευση. Είμαι υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης. Η παράτυπη ε, και παράνομη μετανάστευση ε, είναι, δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει να δούμε και το δικαίωμα του ασύλου, θα δούμε. Δεν έχω με χρόνο τώρα γι' αυτό. Τώρα, για τις αμβλώσεις. Νομίζω ότι οι προσωπικές πεπιθήσεις ε, του καθενός ε, δεν έχουν σχέση με τη δουλειά του. Πάντως, η άμβλωση είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Οπότε, η προσωπική μου άποψη δεν έχει σημασία εδώ. Είναι άσχετη με το έργο που θα αναλάβω, με το χαρτοφυλάκιό μου. Και αν σας ενδιαφέρει, στην Κροατία, την πατρίδα μου, η άμβλωση είναι νόμιμη. Και μάλιστα ήμουν υπέρμαχος στην πατρίδα μου της ε, κύρωσης της σύμβασης της Κωνσταντίνου Και γι' αυτό έχασα και ψήφους συντηρητικών. Γιατί ήμουν ανέκαθεν κατά της βίας της βάρος των γυναικών και της ενδοικογενειακής βίας και το διατράνωσα αυτό στην πατρίδα μου και ήμουν υπέρ τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολεω και ψήφισε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κύρωσή τη. Δεν έχετε κανένα λόγο να αμφιβάλλετε για τι μελλοντικέ μου δραστηριότητε. Ευχαριστώ. Αλεξάνδρα Αλεξάνδρο Γιορτάνοφ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σουίτσα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης. Ο συνάδελφος Κόρμπετ είπε κάτι σχετικό. Ότι δηλαδή υπάρχουν αρχηγοί κρατών που δικαιολογούν την έλευση επιτυχίας τους μέσω, ε, των αποφα... λόγω των αποφάσεων των Βρυξελών. Θα πρέπει πιστεύω να ξεπεράσουμε αυτό το φαινόμενο. Η... Δηλαδή οι κατηγορίες πάντοτε να βαραίνουν τις Βρυξέλλες. Μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα ώστε οι εθνικοί πολιτικοί να σταματήσουν να κατηγορούν διαρκώς τις Βρυξέλλες και να παίζουν πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των Βρυξελών. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ κύριε Γιουρντάνευ για αυτή σας την ερώτηση. Αν θυμάμαι καλά, ε, έγινε μια άτυπη συνεδρίαση των, ε, στο ΣΥΜΠΙΟΥ των, ε, των 27 αρχηγών κρατών και, και, και κυβερνήσεων. Και σε εκείνη τη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα του πώς συμπεριφέρονται οι ηγέτες όταν είναι στη χώρα τους και όταν, πώς όταν είναι στις Βρυξέλλες. Εγώ είμαι κατά των όσων κατηγορούν τις Βρυξέλλες για όλα τα στραβά και μόλις έρχονται στις Βρυξέλλες ζητούν χρηματοδότηση. Δηλαδή τα λεφτά είναι εντάξει, αλλά οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ όχι. Εγώ είμαι εντελώ κατά αυτή τη συμπεριφορά. Είμαι υπερευρωπαίστρια και δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια συμπεριφορά. Έγινε μεγάλη συζήτηση λοιπόν μεταξύ τους τότε και αυτό έγινε γνωστό. Νομίζω πως ο κάθε πολιτικός πρέπει να είναι ανοιχτός και ειλικρινής προς τους πολίτες, να λέει τι ακριβώς είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτή είναι η θέση μου. Да. Ε, ε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας θα έλεγα, θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου, δεν είναι ερώτηση. Η Ένωση θα έχει μέλλον όταν οι πολίτες αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα σταματήσουν να κλέγουν ε, λαϊκιστές για ηγέτες. Πιστεύω πως ε, αν κάτι τέτοιο συμβεί θα είμαστε σαν τις, ε, τη Μεγάλη Βρετανία και τους ηγέτες της. Θα μιλήσω τώρα τη μητρική μου γλώσσα, τα κροατικά, γιατί δεν με έχετε ακούσει ακόμη να μιλάω κροατικά και μια και μιλούμε για πολυμορφία, προτιμώ να απαντήσω στα κροατικά. Τη μητρική μου γλώσσα που είναι η 24η γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν υπάρχει στον κατάλογο κανένας Κροάτης για να θέσει ερώτηση. Θα σας μιλήσω εγώ κροατικά. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συμφωνώ απόλυτα ότι τέτοια πολιτική θα μπορούσε να μας οδηγήσει ε, σε ένα σενάριο όπως αυτό που εξελίσσεται τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντα ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Πάντως τέτοιου είδους λαϊκιστικές, δημαγωγικές δηλώσεις και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν μερικοί να προσετεριστούν τους ε, ψηφοφόρους ή να ε, έχουν μόνο τους στόχο την ψηφοθυρία ε, δεν είναι σωστό. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Οχένια Παλόπ από την Επιτροπή Γυναικών και την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ. Κυρία Σούιτσα, στην Ευρώπη υπάρχουν γυναίκες που θα ήθελαν να έχουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν, γιατί έχουν οικονομικές δυσκολίες, προβλήματα για να συμφιλιώσουν και ε, εμπόδια για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Επίση, στην Ευρώπη υπάρχουν γυναίκε που δεν θέλουν παιδιά και αναγκάζονται να το κάνουν γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε αντισυλληπτικά, δεν μπορούν να κάνουν ε, διακοπή κοίηση. Νομίζω ότι οι γυναίκε έχουμε δικαίωμα να αποφασίσουμε για τη μητρότητα, για, για ε, Και αυτό είναι στοιχείο της δημογραφικής πολιτικής. Πώς θα απαντήσουν οι υπηρεσίες υγείας στο δικαίωμα των γυναικών που έχουν δυσκολίες να αποκτήσουν παιδιά και εκείνων που δεν θέλουν παιδιά και τους υποχρεώνουν, τις υποχρεώνουν για τα παιδιά. Τι λέτε για τις επεμβάσεις ε, που γίνονται στα μεσοφιλικά παιδιά σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τους επιβάλλουν ένα φύλλο, χωρίς να είναι ιατρικά απαραίτητες. Τα δικαιώματα αυτών των παιδιών εσείς πώς θα τα υπερασπιστείτε. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα αυτό. Ε, είναι της Επιτρόπου Υγείας και της Επιτρόπου Ισότητας. Θα συνεργαστώ μαζί τους όμως πάρα πολύ στενά και με τις δύο για να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις. Φυσικά θα πρέπει να προστατεύουμε όλο τον κόσμο, χωρίς διακρίσεις όπως είπατε, όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσπαθούμε να τους βοηθούμε, είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται ε, για τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων ή για άλλες δυσκολίες. Θα συνεργαστούμε και πιστεύω ότι θα βρούμε κάποιες απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις από κοινού. Τώρα δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένη, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Δεύτερη ερώτηση πραγματική, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημογραφία, γι' αυτό σας ρώτησα. Είναι ανησυχητικές οι εξελίξεις στη δημογραφία στην Ευρώπη. Ορισμένοι ε, ανησυχούν από τη μετανάστευση, τις γεννήσεις που είναι κάτω της ανανέωσης και ανησυχούν ότι γερνάνε οι λαοί και τα έθνη και ζουν λιγότερο. Ορισμένοι πολιτικοί υπερσυντηρητικοί της δεξιάς ή της ακροδεξιάς έχουν την πρόθεση να αυξήσουν το δίκτυο των γεννήσεων στην Ευρώπη ε, ποντάροντας στην ετεροφιλοφιλική οικογένεια, την πατραρχική οικογένεια. Αυτό είναι και κατά της οικογένειας και ξενοφοβικό και ομοφοβικό και ε, εισάγει διακρίσεις που δεν συνάδουν με τη συνθήκη. Ε, πώς αντιδράτε εσείς συγκεκριμένα σε αυτά. Στηρίζετε τις δημογραφικές πολιτικές της ακροδεξιάς ε, στη ε, Διεθνή Σύνοδο για τη Δημογραφία που έγινε πρόσφατα στη Βουδαπέστη. Thank Σας ευχαριστώ για τη συμπληρωματική σας ερώτηση. Καταρχάς, εγώ δεν θα χρωματιστώ κομματικά για να σας πω αν υποστηρίζω την ακροδεξιά ή την ακροαριστερά. Εγώ το βλέπω από άλλο πρίσμα. Και πιστεύω ότι η οικογένεια ή οι οικογένειες θα πρέπει, ε, θα μπορούσαν ή οφείλουν να ορίζονται με διαφορετικό τρόπο. Βεβαίω υπάρχει η παραδοσιακή οικογένεια, αλλά δεν είναι ο μόνος τύπος οικογένειας. Ο ορισμός της οικογένειας όμως είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να ε, ορίσω την οικογένεια διαφορετικά, πιο προοδευτικά και πιο φιλελεύθερα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Μπορούμε να συνεργαστούμε. Ανέκαθεν ήμουν πολύ στρατευμένη σε αυτά τα θέματα. Και ακόμα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. Είμαι αντιπρόεδρο των γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και είμαστε πιο προοδευτικέ από όσο ίσω να νομίζετε. Μπονιφέη. Ο κύριος Μπονιφέη για την επόμενη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κυρία Σουίτσα. Η ερώτησή μου αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής δράσης. Δεσμεύεστε, θέλω να σας ρωτήσω, να συμπεριλάβετε στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, στη συνέλευση, μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να εργαστούμε νέα κοινωνικά δικαιώματα που να είναι εφαρμοστέα και ε, να απαιτείται από τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές να τα εφαρμόσουν ε, και έπειτα έτσι να μπορέσουμε να τα μετατρέψουμε σε μια πραγματική κοινωνική χάρτα που να είναι δεσμευτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς σκοπεύετε να στον στηρίξετε αυτό το στόχο. Πώς βλέπετε τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτό το θέμα του πυλώνα και της δημογραφίας που έχετε στο τίτλο του χαρτοφυλακίου σας. Πώς βλέπετε το θέμα των δημογραφικών πιέσεων. Ο πυλώνας εξάλλου θεσπίζει τη βοήθεια, ως άξονα τη βοήθεια για τα παιδιά. Εσείς μιλήσατε για την εγγύηση για τα παιδιά. Χρειαζόμαστε νέο νομικό μέσο και ε, νέο μέσο ε, που να ανέρχεται στα 6 δις ευρώ. Εσείς ε, θα στηρίξετε την ε, χρηματοδότηση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Βονιφέ για την ερώτηση. Μιλήσατε για δεσμευτικό μέσο, μα ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Πυλώνας είναι υποχρεωτικός, απλώς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Θα πρέπει να τον υλοποιήσουμε και αυτό θα μεριμνήσω την ε, υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα. Έτσι αντιλαμβάνομαι την αποστολή μου. Με ρωτήσατε για την εγγύηση για τα παιδιά και την προστασία των παιδιών. Πρόκειται για λιμένη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ενισχυμένο, που προβλέπει 5,9 δισεκατομμύρια. Αυτό ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, για την προστασία των παιδιών και την εγγύηση για τα παιδιά. Εγώ θα είμαι υπέρ και θα ζητήσω και περισσότερα γίνεται. Αλλά ο Επίτροπος Χάν είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, οπότε αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε. Πάντως ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και φυσικά θα λαμβάνω υπόψη ε, τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και είμαι ακόμη εδώ. Κύριε Μπενιφέ, θέλετε να προσθέσετε κάποια άλλη παρατήρηση. Μάλιστα, ευχαριστώ και ευχαριστώ για την απάντησή σα. Βεβαίω το γνωρίζω, γιατί είμαι ένα από του σκιώδει συντάκτε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είμαι ευτυχή ε, για αυτήν την έμφαση που δίνετε για του πόρου. Εσεί θα έχετε ένα χαρτοφυλάκιο πολύ ευρύ ε, για τα θέματα για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, πώ θα ενισχυθεί η δημοκρατία μα, για το θέμα των δικαιωμάτων. Αναφέρ... Ε, ε, ακούστηκαν αμφιβολίες και σε αυτή την ακρόαση για τη δική σας θέση. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω κάποιες συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Σκοπεύετε να δεσμευτείτε στον τομέα της ισότητας των φύλων και ιδιαίτερα το θέμα της ανισο... μισολογικής ανισότητας μεταξύ των φύλων και με ποιο τρόπο. Συμφωνείτε πως η συμφιλίωση εργασιακής με προσωπική ζωή ξεπερνά το απλά το, το, το θέμα της οικογενειακής ζωής και έπειτα για τα δικαιώματα των ανθρώπων που είναι ΛΟΑΔΜΑ. Ε, εσείς ε, πώς θα προωθήσετε το σεβασμό τους στη κοινωνία και στους χώρους εργασίας. Ευχαριστώ για την επερώτηση. Ως Ευρωβουλευτής ε, διατέλεσα και αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΑΦΕΤ και ήμουν μέλος της ε, Επιτροπές Περιβάλλοντος και Γυναικών και είχα ασχοληθεί, ήμουν αρμόδια για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και η δική σας Επιτροπή ε, επίσης λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Οπότε μην ανησυχείτε γι' αυτό. Το θέμα μου είναι προσφυλές και θα το φροντίζω γενικώ και όταν μιλούμε για το χάσμα μεταξύ των φύλων. Γνωρίζετε ότι έχουμε 15% πτυχιούχων α, ανωτά των σχολών γυναικών περισσότερους ε, από άντρες, ενώ 16% ε, έχουμε λιγότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας από άντρες, ενώ είναι πολλαπλάσιος ο αριθμός των γυναικών πτυχιούχων. Ε, εξακολουθούμε λοιπόν να έχουμε μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θα προσπαθήσω να το φροντίσω και αυτό σε Επίτροπος. Πάντως, σε συνεργασία με την Επίτροπο Ισότητας και με τους άλλους Επιτρόπους ή Αντιπροέδρος. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μπορούμε να κατευθύνουμε τα πράγματα και να διαπιστώνουμε την κατάσταση κάθε εξάμεινο. Πολύ σημαντικό εργαλείο. Για τους ΛΟΑΤΚΙ δεν υπάρχει κανένας λόγος διάκρισης ε, εις βάρος οποιοδήποτε. Η απαγόρευση των διακρίσεων είναι ακρογωνιαίος λήθος κατά τη γνώμη μου, οπότε με μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Now, Mrs. Και τώρα... Και τώρα, η κυρία ε, και τη μέλος της Επιτροπής Γυναικών. Ε, Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Κυρία Σουίτσα, στις συνθήκες, όπως γνωρίζουμε όλοι, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να καθορίζονται από πολυμορφία, ε, έλλειψη διακρίσεων, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργαστήκατε και καταψηφίσατε τα δικαιώματα των γυναικών. Καταψηφίσατε το δικαίωμα στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Μπορείτε να, μπορεί να κατηγορείτε άλλους τώρα, αλλά η ψήφωση ήταν αρνητική. Και το να συνδέουμε τις δημογραφικές αλλαγές με το ε, δικαίωμα επιλογής των γυναικών να αποφασίζουν για το σώμα τους είναι ο κρογονέος λήθος των πολεμίων της, των αυλώσεων παγκοσμίω. Στις δημοκρατίες μια ασφαλής πρόσβαση στην αύλωση είναι δικαίωμα ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιώδων ελευθεριών και όχι μόνο θέμα δημοκρατίας. Θα μας Μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι θα προωθήσετε τα δικαιώματα των γυναικών να αποφασίζουν για το κορμί τους και για την σεξουαλικότητά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κούνκε. Ξέρω ότι ήσασταν και υπουργό στη Σουηδική κυβέρνηση με αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Να διευκρινίσω την ψήφα μου, γιατί έχω ακούσει παρελειμμένως αυτό το επιχείρημα ότι ήμουν κατά των δικαιωμάτων των γυναικών. Θυμάστε την έκθεση Ζούμπερ και την έκθεση Εστρέλα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η πρώτη χρονιά που χάρισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν το 2013-2014, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν η πρώτη μου θητεία που κράτησε μόνο ένα χρόνο, γιατί το 2013 η Κροατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ναι, ψήφισα κατά. Ψήφισα κατά όχι γιατί είμαι κατά των δικαιωμάτων των γυναικών ή ήμουν κατά της ισότητας των φίλων, Ψήφισα κατά γιατί οι δύο εκθέσεις περιλάβαναν στοιχεία που ήταν τελείως άσχετα με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Και οι δύο εκθέσεις, και η έκθεση Ζούμπερ και η έκθεση Εστρέλα, αν θυμάστε, δεν είχαν τελικά εγκριθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπερψηφίστηκαν γιατί ζητούσαν επιπλέον δημοσιονομικούς πόρους και τότε ήμασταν ακόμη εν μέσω της κρίσης. Και δεν υπήρχε συνένεση ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπερψηφιστούν οι δύο εκθέσεις. Και αυτό ήταν ένα από του λόγου που καταψήφισα τις δύο εκθέσει. Και σε μία από αυτέ δεν θυμάμαι αν ήταν η έκθεση Ζούμπερ ή η έκθεση Εστρέλα, ε, είχα καταθέσει, είχαμε, είχε καταθέσει η πολιτική μου ομάδα ένα εναλλακτικό ψήφισμα. Και είπα στην αρχή, καλύτερα να προέρχεται κανείς από ένα περιφερειακό ή ένα εθνικό κοινοβούλιο και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τη στιγμή που είναι κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φυσικά πολιτικός είναι και προσπαθεί να σταθμίσει τις πολιτικές του απόψεις, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είμαι ουδέτερη. Και γι' αυτό προσπαθώ να εξηγήσω αυτό το ιστορικό μου στις ψηφοφορίες και το πώς ψήφισε σε μερικές εκθέσεις. Κυρία Σουίτσα, ναι, ακούω τις απαντήσεις, αλλά δεν απαντήσατε σε αυτό που σας ρώτησα για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Εσείς, βάσει των συνθήκων, θα υπερασπίσετε και θα προωθήσετε τα δικαιώματα αυτά για όλους. Θα προωθήσετε και θα υπερασπίσετε και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Θα προασπίσετε και θα προωθήσετε τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των προσφύγων για παράδειγμα. Θα υπερασπίσετε τα δικαιώματα των Εβραίων και των Μουσουλμάνων. Θα υπερασπίσετε τα δικαιώματα των γυναικών να αποφασίζουν για τη σεξουαλικότητα και το σώμα τους. Ευχαριστώ για την επερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προτείνω είναι τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτου δικαίου, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτέ είναι οι αξίε που είναι κοινέ ε, ε, σε μια κοινωνία που η πολυμορφία, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη και η ισότητα ανδρών και γυναικών πριτανεύουν. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλω, όπως προβλέπει και την κατοχυρώνει και το άρθρο 2. Και αυτό θα το τηρώ πάντα. Μείνετε ήσυχοι λοιπόν και μην αμφιβάλλετε για τις πεπιθήσεις μου, ούτε για τις μελλοντικέ μου δραστηριότητες ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Γιάννα Τόμ από την ομάδα Renew Europe, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ξέρω ότι δεν είναι του χαρτοφυλακίου σας, αλλά ειλικρινά δεν έχω καταλάβει τα χαρτοφυλάκια ακριβώς και πού εντάσσετε. Πανελημέρα μιλήσατε για το κοινωνικό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων ως ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά είπατε επίσης ότι είναι στα κράτη-μέλη, στα χέρια τους με βάση την επικορικότητα. Ισχύει αυτό. Απαντώντας σε κάποια ερώτηση, είπατε ότι ένας καλός τρόπος να δείσουμε στα κράτη-μέλη πώς θα πρέπει να δράσουν είναι οι συστάσεις αναχώρα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εδώ από τους 18 που μίλησαν, μόνο τρεις είναι μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης. Από το 2012 μέχρι το 2018 μειώθηκε σημαντικά η εφαρμογή των συστάσεων από τα κράτη-μέλη. Από το 72% έπεσε στο 39%. Και μάλιστα ήταν ελλειπής η εφαρμογή. Ε, υπήρξε κάποια πρόοδο στο, πέρυσι στο 39% των συστάσεων και όχι πλήρη εφαρμογή. Πώς θα αναγκάσετε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αυτές τις ε, συστάσεις Αλλιώς μετά από πέντε χρόνια θα μιλάμε 18% που επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος. Ε, πώς θα λυθούν τα προβλήματα που είναι δική σας αρμοδιότητα. Κατανοώ την ερώτησή σας και σας ευχαριστώ. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Γιατί αν τα κράτη-μέλη δεν ακολουθούν τις συστάσεις, τότε τι να το κάνουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Πολύ καλή ερώτηση. Είπατε ότι δεν είναι το δικό μου χαρτοφυλακίου, αλλά είναι μία από τις ευθύνες που έχω γιατί θα συνεργαστούμε και ε, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να χειραφετήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη για να τηρούν τις συστάσεις. Σίγουρα θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και θα φροντίσουμε τα κράτη-μέλη ε, να δρούν σύμφωνα με τις συστάσεις που τους απευθύνονται διαφορετικά να το καταργήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό όμως είναι μια ερώτηση για την κυρία Φόντερ Λάιεν ή για τον κύριο Ντομπρόφσκης που είναι αυτό το διάστημα στο χαρτοφυλάκιό του. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και είναι ίσως το μοναδικό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δράσει και να προκαλέσει την αντίδραση των κρατών μελών στις συστάσεις. Όχι μόνο σε αυτό το τομέα, αλλά σε πολλούς τομείς όπως γνωρίζουμε. Αλλιώς προσφεύγουμε στο δικαστήριο. Και άμα αρχίσει στα δικαστήρια είναι ε, μακρές οι διαδικασίες μετά τα πρόστιμα και δεν είναι προς το συμφέρον κανενός κράτους μέλους. Ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλωστε. Παρακαλώ, συμπραγματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πρώην δημοσιογράφος και δεν πιστεύω ε, σε ε, παραθέσεις. Ε, προηγουμένως είπατε στον συνάδελφο Μπενιφέη ότι ο κοινωνικός πυλώνας είναι δεσμευτικός για τα κράτη-μέλη. Σωστά σας παραθέτω λέγοντας ότι η άμβλος είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ως μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή θα ανεχτείτε τα κράτη-μέλη ε, που νομοθετούν για να απαγορεύουν τις αμβλώσεις. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αυτό που είπα, να το εξηγήσω. Είναι, να σας εξηγήσω τι γίνεται με την άμβλωση. Η άμβλωση, όπως είπα, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Υπάρχουν νομοθεσίες, στη χώρα μου επιτρέπεται, σε άλλες χώρες απαγορεύεται η άμβλωση, αλλά σύμφωνα με το συλλογικό πνεύμα της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εργαστώ προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό σας είπα. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό πυλώνα, γνωρίζω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα. Το δεσμευτικό ήταν εντός εισαγωγικών όταν το είπα. Δηλαδή, καλό θα ήταν αν τα κράτη-μέλη ε, τηρούσαν τον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα. Γιατί, ε, δεν ξέρω, συγγνώμη αν παρεξηγήθηκα, δεν το διατύπωσα σωστά. Δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί παρεξήγηση, δεν νοούσα κάτι διαφορετικό ή κάτι αντίθετο με αυτό. Και τώρα, ο κύριος Κονθάλης Πόνς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Καλησπέρα σα, ε, κυρία υποψήφια Επίτροπε. Εγώ είμαι μέλο τη Επιτροπή ε, Γιούρι και θέλω να ε, πω στου συναδέλφου πω η υπόθεσή σα πέρασε χωρί καμία συζήτηση. Όταν η Επιτροπή Γιούρι συζήτησε για το ποιο επίτροπο μπορούσε να έχει ε, σύγκρουση συμφερόντων και ποιο όχι. Εσείς ήσασταν σε εκείνους που δεν είχαν σύγκρουση συμφερόντων. Έχω δει το βιογραφικό σας και ξέρω πως έχετε εμπειρία, αλλά όχι μόνο επειδή ε, σας ξέρω γιατί ήσασταν μαζί μας, ψηφίζατε μαζί με το ΕΛ και κάθε φορά που σας, επικρίνουν για τις προηγούμενες σας θέσεις, επικρίνουν ολόκληρο το ΕΛΚ, ολόκληρο το Λαϊκό Κόμμα, γιατί εκείνη πάντοτε ψήφιζε το ίδιο με ό,τι ψηφίζαμε οι υπόλοιποι. Εγώ δεν πιστεύω στο ένα κοινοβούλιο στο οποίο όλοι ψηφίζουν το ίδιο. Ούτε ένα κοινοβούλιο που λογοκρίνονται τα μέλη του επειδή ψήφισαν όπως ψήφισαν. Πιστεύω ένα κοινοβούλιο όπου ο καθένας έχει την ελευθερία να ψηφίζει αυτό που πιστεύει. Εμείς ε, ψηφίσαμε μαζί με την Επίτροπο. Είμαστε το γκρουπ, η ομάδα που έχει την πλειοψηφία σε αυτό το σώμα. Επειδή ακολούθησε μια γραμμή ψηφοφορία, ε, δεν μπορεί να λογοκριθεί. Ε, δεν μπορείτε να μας κατακρίνετε ολόκληρο την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επειδή ψηφίσαμε όπως ψηφίσαμε. Τώρα, αν κάθε φορά που σας ζητάμε θα έρχεστε ή είστε μόνο εδώ επειδή είστε υποχρεωμένοι για την ακρόαση και τι έχετε να πείτε για το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ κύριε Γκονζάλες Πόνς. Αυτό ήμουν έτοιμη να πω. Σκεφτόμουν ότι αν δεν ήμουν μέλος του Ευρωκοινοβουλίου θα ήταν δύσκολο να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά, γιατί είναι πολύ περίπλοκο το χαρτοφυλάκιο. Αν δεν παρακολουθούσα δηλαδή τα όλα όσα κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και τώρα βλέπω πως το να είμαι ευρωβουλευτής είναι ε, μειονέκτημα. Εγώ σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ε, εντάξει, κάποιες φορές υπήρχε και ελεύθερη ψήφος και αποφάσιζα μόνη μου. Κάποιες άλλες φορές, ναι, ακολουθούσα τη γραμμή της ομάδας μου. Σας ευχαριστώ. Αλλά άσχετα από όλα αυτά, είδα ότι αυτή η Επιτροπή, όχι η Επιτροπή Απασχόλησης, ούτε η Επιτροπή Γυναικών, αλλά η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ε, ε, είχαμε και ασχοληθήκαμε με τις σωστές πρωτοβουλίες για πολλά πολλά χρόνια και αυτό ε, το βλέπουμε σε όλες τις εκθέσεις. Όμως, εξεκολουθούμε να έχουμε κάποια πρωτοβουλία σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά όπως ε, λέγεται και στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές ε, από πλευράς της ε, υποψήφιας Πρόεδρου, εκείνη το επιθυμεί, θα το επιθυμώ και εγώ να αλλάξουμε τα πράγματα και να δώσουμε δικαίωμα πρωτοβουλία αν αυτό το ε, αποφασιστεί. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτή που θα το αποφασίσει σήμερα. Δεν θα το καταψηφίσω. Είμαι από, ε, προέρχομαι από το Κοινοβούλιο και θέλω να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του και ξέρω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Θα έρθω λοιπόν, θα το συζητήσουμε και θα δούμε πώς θα, θα, θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ε, κύριε Γκοζάλες Πόνς, ναι, θα ήθελα να αναφέρω μια έκθεση, την έκθεση Γκοζάλες Πόνς για τους καντιντάτ. Το αναφέρω ως υπεύθυνο για την έκθεση αυτή, αλλά και ως μέλος του ΕΛΚ. Θα μιλήσουμε για το θεσμό των καντιντάτ. Έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό ή να πούμε ότι έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση και ότι η έκθεσή μου θα ξεχαστεί για πάντα. Αγαπητέ Στεμπαν, δεν έχει τελειώσει και δεν θα ξεχαστεί και στην, επιστολή ανάθεση της εντολής ε, ε, και σε άλλων ε, συναδέλφων ε, αναφέρεται ότι πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη και ότι πρέπει να συζητηθεί. Θα είναι το πρώτο θέμα στη, για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Η Spitzenkandidat και η, η τα διακρατικά ψηφοδέλτια. Ε, πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την υπόθεση γιατί, γιατί θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να καταλάβουν τι συμβαίνει. Διαφορετικά ε, τους έρχεται λίγους μήνες πριν από τις και δεν ξέρουν να κάνουν. Είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή τη φορά απέτυχε, αλλά εγώ πιστεύω πως είναι καλό το σύστημα αυτό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ξέρουν για ποιον ψηφίζουν και πιστεύω πως ε, η ισχύ των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα είναι πολύ σημαντική. Γιατί τότε θα έχουν ε, εκεί λόγο. Περισσότερο από ό,τι έχουν τώρα. Μέχρι τα τέλη του επόμενου καλοκαιριού, λοιπόν, όπως υποσχέθηκε η υποψηφία πρόεδρος, θα το έχουμε ε, συζητήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκοζάλες Πόνς. Ήταν αυτή η τελευταία ερώτηση από πλευράς των ε, Ευρωβουλευτών ε, τώρα. Η υποψήφια αντιπρόεδρος έχει πέντε λεπτά για να προβεί στις τελευταίες της παρατηρήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμε πρόεδρε και αγαπητά μέλη, έχω προετοιμάσει ομιλία, αλλά δεν πρόκειται να τη διαβάσω. Νομίζω καλύτερα να σας μιλήσω απευθείας απ' έξω. Νομίζω ότι η, η συζήτηση αυτή ήταν πολύ καλή, γόνιμη, συναρπαστική, έντονη για μένα, αλλά και πολύ χρήσιμη, γιατί διαπίστωσα την πολυμορφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την πολυφωνία, την ποικιλία απόψεων και αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για το μελλοντικό μου έργο, εφόσον φυσικά με εγκρίνεται για την ε, ανάληψη των καθηκόντων μου. Πάντως θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα βάλω τα δυνατά μου στο χαρτοφυλάκιό μου για να γίνει το χαρτοφυλάκιο ε, Δημοκρατία και Δημογραφία ένα χαρτοφυλάκιο που θα πλησιάσει τους πολίτες και το πιο σημαντικό ε, είναι η γύρανση, η συμφιλίωση επαγγελματικού και προσωπικού βίου και τα παιδιά. Δηλαδή όλο το σύνολο της ζωής με επίκεντρο το πολίτη. Αυτό θα είναι το χαρτοφυλάκιό μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πάντα μιλάμε ότι θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική η πολιτική μας, να έχει στην καρδιά της τον πολίτη. Και αυτό θα είναι το μέλημά μου την επόμενη πενταετία αν πάρω την έγκρισή σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τη συζήτηση που είχαμε. Όπως είπα και στην αρχή, ήμουν μέλος σε πολλές επιτροπές και προσπάθησα να το λάβω αυτό υπόψη στην προετοιμασία μου, γιατί αφιέρωσα αρκετές εβδομάδες στην προετοιμασία αυτή. Όταν συνειδητοποίησα ότι θα αναλάβω αυτό το χαρτοφυλάκιο, άρχισα να μαθαίνω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα για να προετοιμαστώ, για να κατατοπιστώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν θέμα αρμοδιότητάς μου. Ήμουν περισσότερο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ή ήμουν πιο κοντά στους πράσινους, στη στρατηγική για κατά των πλαστικών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παρόλο που με διέφεραν και τα θέματα του χαρτοφυλακίου μου, αλλά όχι τότε άμεσα άλλα συστήματα παρακολουθούσα ως Ευρωβουλευτής και μέλος διαφόρων επιτροπών. Και αναπτύσσοντας αυτό το χαρτοφυλάκιο θα χρησιμοποιήσω τρία εργαλεία. Την εδραίωση, την επικοινωνία και την επικοινωνία. Επικοινωνία, εμπέδωση και συνεργασία. Αυτά θα είναι τα τρία αυτές τις τρεις κατευθυντήρες γραμμές της ε, πολιτικής μου. Θέλω επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μη κυβερνητικέ οργανώσει, κοινωνία των πολιτών, τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Και σα είπα και στι γραπτέ μου απαντήσει ότι για 10 χρόνια ήμουν στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, αντιπρόεδρο ε, του Συνεδρίου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Αυτή ήταν η θέση μου, γιατί ήμουν δήμαρχος του, στο Ντούμπροβνικ, οπότε και 10 χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο της Ευρώπης και παρακολούθησα στενά τα τοπικά και περιφερειακά ζητήματα. Οπότε το θέμα της συνεργασίας είναι πολύ σημαντικό, της εδραίωσης, αλλά και της επικοινωνίας. Επικοινωνία με τους πολίτες, με το κοινό, ε, θα πρέπει να φτάσουμε στον πολίτη, να τον αγγίξουμε, να τον πλησιάσουμε και όχι να μείνουμε ε, οχυρωμένοι στις Βρυξέλλες, στη φούσκα των Βρυξελών. Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε αποξερωμένοι στον κόσμο μας, αλλά να φτάσουμε στις, ε, στους πολίτες στις πιο απόμακρες περιοχές, στην κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και τώρα να ρίξω και μια ματιά στις σημειώσεις μου. Και να σας πω εν το εξής. Γνωρίζετε ότι κατάγομαι από μια χώρα και έγινα μάρτυρας, είδα με τα μάτια μου την πατρίδα μου να εκδημοκρατίζεται, να ανακτά την ανεξαρτησία της και να γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια διαδικασία που κράτησε περίπου μια τριακονταετία και ήμουν αυτόπτης μάρτυρας όλης αυτής της διαδικασίας. Τώρα είμαστε και εμείς μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας και είμαστε πανευτυχείς γι' αυτό. Και γι' αυτό αυτή την εμπειρία μου θα τη μεταφέρω και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, γιατί κάποιος με ρώτησε για τις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Θα τις βοηθήσω να προετοιμαστούν για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί νομίζω ότι όλοι προσβλέπουν να ενταχθούν σε αυτή την φημισμένη λέσχη. Λυπάμαι ε, για μερικούς είναι πια πολύ αργά γιατί αποφάσισαν να φύγουν, αλλά νομίζω ότι πολλοί θα ήθελαν να ε, ενταχθούν σε, αυτή αυτό τη λέσχη που έχει τόσο κύρος. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την συζήτηση και την αξιολόγηση και θα είμαι συνάδελφός σας, ακόμη και γίνονται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ε, αν γίνω αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώ. Η δεμή θα παραμείνω συνάδελφό σα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Υποψήφια Αντιπρόεδρε, για τις απαντήσεις σας και για την δέσμευση σας ειδικά όσον αφορά την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν σε αυτή την ακρόαση. Ευχαριστώ φυσικά και τους διερμηνείς που μας επιτρέψατε να μιλήσουμε όπως εγώ τώρα στις μητρικές μας γλώσσες. Σας θυμίζω ότι οι συντονιστές θα, για θα συνεδριάσουν στις 22 και 30 και κλεισμένων των θυρών για την αξιολόγηση και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές το έβδομο ε, ε, παράρτημα του κανονισμού της, ε, του Κοινοβουλίου ορίζει ότι σκοπός της ακρόσης είναι να δούμε την ευρωπαϊκή προσήλωση για την προσωπική ανεξαρτησία καθώς και τις γνώσεις του για το μελλοντικό του καθορτοφυλόγιο καθώς και τις δυνατότητες της επικοινωνιακές του. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η απόψηνή ακρόαση. Ευχαριστώ.